Bueno, buenos días. Καλημέρα σα. Να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την ημερήσια διάταξη. Καταρχάς, Σημείο 2. Έγκριση της μερίσιας διάταξης. Να σας πω ότι έχει γίνει μια αλλαγή στο σημείο 10 ψηφοφορία για το Ανασύσταση του αποθέματο του Ευρωπαϊκού Χελιού αναβάλλεται για την επόμενη συνεδρίαση, καθώς επίσης και το στρατηγική για την ε, Αδριατική και το Ιόνιο Πέλαγος. Τα δύο αυτά σημεία δηλαδή, σημεία 10 και 11, δεν θα ψηφιστούν σε αυτή τη συνεδρίαση. Δεν υπάρχει κάποια άλλη αλλαγή. Συμφωνείτε με αυτές τις αλλαγές. Ωραία λοιπόν. Περνάμε τώρα στην έγκριση των πρακτικών της συνεδρίασης της 22ης και 23ης Απριλίου. Θα είδατε ότι τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης ε, σας είχα ενημερώσει εν συντομία για τις διαπραγματεύσεις για το βασικό οριζόντιο κανονισμό για την ε, κοινή πολιτική αλληλείας και αυτό δεν συμπεριλήφθη στα πρακτικά. Το λέω λοιπόν για να συμπεριληφθεί στα πρακτικά αυτή η μικρή ενημέρωση που έγινε και οι πληροφορίες που δόθηκαν ε, σε εκείνη τη συνεδρίαση διαφορούν ε, τα ε, του βασικού κανονισμού για την ε, μεταρρύθμιση κοινή ελευτικής πολιτικής. Αν δεν υπάρχει κάποια ένσταση μέχρι το πέρας της συνεδρίασης θα θεωρούμε ότι εγκρίνονται τα πρακτικά. Τώρα, για τις ανακοινώσεις του Προέδρου πρέπει να σας πω ότι για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και ο κύριος Καντέκ προτείνει μια νέα προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών για τα άρθρα τα οποία τροποποιήθηκαν, δηλαδή τα άρθρα 94 έως 107 και ζητά να δοθεί προθεσμία για τις ε, τροπολογίες μέχρι την 5η 6 Ιουνίου. Μέχρι τότε λοιπόν θα μπορείτε να καταθέσετε τροπολογίες. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αλλάξει το χρονοδιάγραμμα. Θα παραμείνει ως έχει και η ψηφοφορία θα γίνει ε, όπως προβλέπετε για τις 10 Ιουλίου. Me indican que, que en Από ό,τι φαίνεται, σε αυτή την περίπτωση δεν θα μπορέσετε να κατεθέσετε τροπολογίες ε, με το... ή μάλλον διορθώνει ο πρόεδρος, πρέπει να τη στείλετε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και όχι με το αυτόματο σύστημα ε, υποβολής τροπολογιών. Ερωτήσεις? Όχι, ωραία, να περάσουμε στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης για μια ολοκληρωμένη ελευθερική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή του Ειρηνικού. Σήμερα θα γίνει μια πρώτη ανταλλαγή απόψεων με την εισηγήτρια, την κυρία Φράγα, στην οποία δίνω και αμέσω το λόγο. Ναι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχάς θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη διότι παρά το γεγονός ότι μου ανατέθηκε αυτή η έκθεση εδώ και αρκετό καιρό, επειδή όπως θα σας εξηγήσω ε, υπήρξαν διαπραγματεύσεις και είναι ακόμα να εξελίξει διαπραγματεύσεις εντός του Συμβουλίου με τις χώρες του Ειρηνικού, κυρίως ε, στα πλαίσια της ε, Οικονομικής Συμφωνίας Εταιρικής Σχέσης, καθώς επίσης και διαπραγματεύσεις για την αξιολόγηση των πιθανών συμφωνιών με άλλες χώρες της περιοχής, ε, καθυστέρησε. Ειδικά το θέμα της εταιρική σχέσης είναι πολύ σημαντικό γιατί εκεί περιλαμβάνονται και τα θέματα της αλίας. Οι διαπραγματεύσεις αυτές όπως θα σας εξηγήσω δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα και ήθελα να περιμένω λίγο για να δούμε ποιες θα είναι οι τελικές αποφάσεις για λόγους οι οποίοι δεν είναι της δικής μας αρμοδιότητες, ε, οι πολιτικές ομάδες αποφάσισαν ότι οι εκθέσεις πρωτοβουλίας οι οποίες είναι εν εξελίξει θα πρέπει να προχωρήσουν πιο γρήγορα για κάποιο λόγο που δεν κατανοώ, αλλά ε, αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε συζητήσεις, αλλά θα ήθελα να ξεκινήσουμε και τη συζήτηση για να ακούσω και τις απόψεις σας και να ετοιμάσουμε λίγο την έκθεση ε, και όταν θα έχουμε και τα αποτελέσματα, αν τελειώσουν ποτέ αυτές οι διαπραγματεύσεις, να έχουμε και τα τυχόν αλλαγές ε, στην έκθεση. Για το θέμα αυτό να σας πω ότι ο βασικός στόχος της στρατηγικής για τον ειρηνικό είναι να καθορίσουμε στην περίπτωσή μας μια αλλιευτική στρατηγική μακροπρόθεσμη, αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και ένας καλύτερος συντονισμός όλων των κοινοτικών πολιτικών ε, που εφαρμόζονται στη συγκεκριμένη περιοχή του Ειρηνικού, ώστε να είναι και ε, πολλαπλό το αποτέλεσμα γνωρίζετε νομίζω αρκετοί εδώ, ε, αρκετά πράγματα, ίσως και περισσότερα και από μένα. Η περιοχή του Ειρηνικού είναι ο πιο πλούσιος ε, ωκεανός ε, στα κυρίως μεταναστευτικά είδη. Το μεγαλύτερο τμήμα των θηνοειδών ξεκινούν από εκεί και το 70% των αλλιευμάτων γίνεται στον κεντρικό και δυτικό ειρηνικό. το ξέρω ότι σας τα λέω όλα λίγο συμπούρδουλα εδώ πέρα, αλλά όπως γνωρίζετε αυτή τη στιγμή ε, ετοιμαζόμαστε για την συμφωνία μετά το Κοτονού. Το, η συμφωνία του Κοτονού εκπνέει το 2020 και γι' αυτό και η αλλιευτική στρατηγική σε μακροπρόθεσμο πλαίσιο θα πρέπει λίγο να ε, εστιάσει και στο τι ακριβώς θα γίνει μετά το Κοτονού. Επειδή ακριβώς λοιπόν μελετάμε το τι θα γίνει μετά το Κοτονού, ε, όλα ε, επικεντρώνονται σε περιφερειακό επίπεδο. Έχουμε ένα πλαίσιο σαν αυτό που έχουμε τώρα, χώρες ΑΚΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα δούμε και κατά πόσο θα μπορούσαμε να έχουμε και ε, συμφωνίες σε περιφερειακό επίπεδο. Το περιφερειακό ζήτημα έχει μεγάλη σημασία για το Κοτονού και ε, η δική μας στρατηγική ίσως θα μπορούσε να χρησιμεύσει ώστε να υπάρχει μια κατάλληλη ελιευτική στρατηγική που να μπορεί να βοηθήσει και να έχει κάποιο νόημα σε αυτή την ανάλυση που κάνουμε για το τι θα γίνει μετά το κοτονού μας ενδιαφέρει κυρίως από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης η οικονομική ανάπτυξη. Η οικονομική ανάπτυξη μέσω προσαρμογής στην αλλαγή του κλίματος, μέσω μιας ε, κατάλληλης εμπορικής πολιτικής και ταυτόχρονα ε, βιώσιμης ε, εκμετάλλευσης των αλλιευμάτων μέσω μιας διάφανης διαχείρισης. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία τα οποία θεωρεί στοιχειώδη η Ευρωπαϊκή Ένωση για τη στρατηγική στη συγκεκριμένη περιοχή ε, μετά θα μιλήσω λίγο περισσότερο για την περιοχή του κεντρικού και δυτικού ε, ειρηνικού, όπου βρίσκονται και όλες οι χώρες ΑΚΕ. Και τώρα θα σταθώ σε ένα κυρίως αλλιευτικό ζήτημα. Σε όλο τον ειρηνικό υπάρχουν τρεις περιφερειακούς οργανώσεις αλλίας. Μία εξ αυτών, ή ε, μάλλον οι δύο εξ αυτών είναι οργανώσεις για θηνοειδή και οι άλλοι δεν είναι. Η πρώτη, θα τα πω κατά αρχαιότητα, είναι ε, η οργάνωση του τροπικού τόνου, Αυτή είναι μια περιφερειακή οργάνωση αλληλεία που ασχολείται κυρίως με τα μεταναστευτικά είδη των θηνοειδών και καλύπτει την ε, βασική περιοχή από τον κεντρικό ειρηνικό ε, της Ηνωμένες και τη Χιλή και ε, ασχολείται με τα θηνοειδή στην περιοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μέλο από το 2006 και πλέον διαθέτει ένα στόλο ισπανικό κατά βάση περίπου 30 σκαφών που δραστηριοποιούνται στη συγκεκριμένη περιοχή του Ειρηνικού. Η δεύτερη μεγάλη περιφερειακή οργάνωση Αλίας είναι η οργάνωση Αλίας για τον Δυτικό και Κεντρικό Ειρηνικό, Western and Central Pacific Fisheries Committee, η οποία ασχολείται με την διατήρηση των θηνοειδών και άλλων υψηλά μεταναστευτικών ειδών σε στις περιοχές του κεντρικού και δυτικού ειρηνικού είναι πιο πρόσφατη από την προηγούμενη, διότι συστάθηκε το 2004, είναι πρόσφατη λοιπόν, και αυτή τη στιγμή ο κοινοτικό στόλων ως έχει άδεια αλίας ε, στα πλαίσια της Συμφωνίας Αλίας για τέσσερα ε, ε, τέσσερις γρήπους και επτά παραγαδιάρικα σκάφη. Και η πιο πρόσφατη περιφερειακή οργάνωση αλίας, ε, και μάλιστα νομίζω ότι ήμασταν και όλοι εδώ και εγώ ήμουν και εισηγήτρια για το θέμα αυτό, είναι η περιφερειακή οργάνωση για τον ε, νότιο ειρηνικό που ασχολείται με κυρίως πελαγικά είδη. Το πιο σημαντικό είδος για μας είναι το σκουμπρί και φυσικά υπάρχουν και κάποια άλλα ε, πελαγικά είδη. Το 2012 ολοκληρώθηκε η συμφωνία, κύρωσε και η Χιλή τότε και έχουμε ε, σκάφη τα οποία αλλιεύουν πελαγικά είδη από την Ολλανδία, τη Γερμανία και την Ιρλανδία που ασχολούνται με την αλληλεία αυτών των ειδών που εκπροσωπεί η Περιφερειακή Οργάνωση. Αυτές είναι οι τρεις περιφερειακές οργανώσεις ε, στις οποίες συμμετέχει η Ευρωπαϊκή Ένωση και έχουμε και στόλο σε όλες τις ε, οργανώσεις ε, σχετικά μικρό ε, είναι σημαντικό, αλλά παντού υπάρχει εκπροσώπηση. Όσον αφορά τώρα τις διμερείς συμφωνίες, οι ε, εταιρικέ ε, συμφωνίες αλλιες ε, θα γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι η πιο παλιά είναι η συμφωνία η οποία έχει συναυτεί με το Κυριμπάτι. Μετά υπάρχουν συμφωνίες για τα νησιά του Σολομόντα και τη Μικρονησία με πολλά προβλήματα όπως γνωρίζετε και αυτές τις δύο συμφωνίες. Η συμφωνία της Μικρονησίας δεν έχει αποτελέσματα εδώ και χρόνια παρά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε την πρώτη δόση της οικονομικής ενίσχυσης και μάλιστα και η ήδη οι εφοπλιστές ε, πλήρωσαν για άδειες αλλοίε που δεν ξέρω αν τους έχουν επιστραφεί και τα χρήματα, θα μας τα πει ο διευθυντής που είναι παρόν. Και η συμφωνία με τα νησιά του Σολομόντα έχει σταματήσει γιατί θεωρούν τα νησιά του Σολομόντα τώρα ότι καλύτερα θα ήταν να έχουν ένα άλλο πρόγραμμα το οποίο θα εξηγήσω αργότερα. Ε, το Vessel Deal Scheme, ε, αλλά και εκεί έχουν σταματήσει τα θέματα. Υπάρχουν κάποιες διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή για να αξιολογήσουμε κατά πόσον υπάρχει δυνατότητα να ζητηθεί και κατάλληλη εντολή, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει ζητηθεί εντολή διαπραγμάτευσης από το Συμβούλιο με τα νησιά του Κουκ και με το Τουβάλο, Βάλου. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι σε διαπραγματεύσεις με αυτά τα νησιά και κυρίως νομίζω ότι με τα νησιά Κουκ έχουμε προχωρήσει λίγο περισσότερο από ότι με το Τουβάλου. Τα θέματα αυτά λοιπόν είναι καθαρά λευτικά ζητήματα και νομίζω ότι λίγο πολύ θα πρέπει να γνωρίζουμε όλοι και τώρα θα ήθελα να σας πω και κάποιες σκέψεις μου διότι αυτή η περιοχή είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα από πλευράς λευμάτων και εμπορίου ε, τόνου. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω κάποιες σκέψεις μου για την παγκόσμια αγορά τόνου. Ε, κυρίως ε, δεδομένου ότι μιλάμε για αυτή την περιοχή η οποία ε, έχει πολλά αποθέματα τόνου. Έχω κάποια στοιχεία του 2009 τα οποία τα έχουμε συγκρίνει και με το ΦΑΟ και με άλλα στοιχεία. Τα αλλιεύματα των θηνοειδών είναι λίγο πολύ σταθερά. Είναι 4.400.000 τα μεταναστευτικά είδη, αυτά είναι τα ποσά από 4.200 μέχρι 4.400 και οι περισσότεροι θεωρούν ότι είναι σταθερός αυτός ο αριθμός, δεν θα αυξηθεί, μάλλον θα μειωθεί, αλλά προς το παρόν είναι σταθερός αυτός ο αριθμός. Το 80% του τόνου καταναλώνεται σε κονσέρβα. Επομένως, το εμπόριο της κονσερβοποιίας τόνου είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεδομένου ότι το 80% του τόνου πηγαίνει στην κονσερβοπία. Από αυτές τις κονσέρβες τόνου, την ε, συγκεκριμένη διαδικασία μεταποίησης, το 8% είναι κοινοτική παραγωγή, ενώ το 92% αυτού του 80% είναι παραγωγή τρίτων χωρών. Η μεγάλη όμως μετεγκατάσταση της ε, κονσερβοποίησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να πούμε ότι έχει ήδη γίνει και θα ήταν πολύ δύσκολο να μειωθεί περισσότερο από αυτό το 8% διότι κάπου υπάρχουν τα όρια στη ζωή. Ε, θα μπορούσε ίσως να παράγει περισσότερο, αλλά όταν ε, μας είχε πει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι ε, υπάρχουν μετεγκαταστάσεις στην Ευρωπαϊκή Βιομηχανία που ασχολούνταν με άλλο θέμα βέβαια, το οποίο δεν μας αφορά και δεν θα σχολιάσω εδώ, ε, αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ κοινοτική παραγωγή. Μπορεί να είναι καλή, ποιοτική και ούτω καθεξής, αλλά αυτή είναι. Και επειδή η αγορά του τόνου είναι ε, πολύ ευαίσθητη και ανέκαθεν το θέμα του τόνου ήταν ευαίσθητο, Ισχύει και το γεγονός ότι οποιαδήποτε παραχώρηση, και εδώ αναφέρομαι στην ε, εμπορική πολιτική, ε, οποιαδήποτε παραχώρηση γίνει σε τρίτη χώρα σε εμπορικά ζητήματα έχει συνέπειες και για τους υπολείπους. Επειδή λοιπόν η κοινοτική παραγωγή είναι σταθερή και το μεγαλύτερο τμήμα παράγεται στο εξωτερικό, οποιαδήποτε δασμολογική παραχώρηση κάνουμε εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωσης κυρίως έχει συνέπειες για τις τρίτες χώρες μεταξύ τους. Και αυτό το είδαμε κατά κάποιο τρόπο και στην περίπτωση της Παππούας Νέας Γουινέας, ε, όταν στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου διαπιστώθηκε ότι όλα αυτά είχαν συνέπειες για τους υπολείπους. Θα θυμάστε ότι σε Σεϊχέλες όταν είχαμε πάει στην αντιπροσωπεία εκεί είχαν πει ότι είχαν παρατηρήσει αυτό το θέμα αυτό. Και το λέω εδώ, είναι ίσονο σημασία σε αυτό το ζήτημα. Έχει σημασία περισσότερο για το Βιετνάμ που είναι η πιο ανταγωνιστική χώρα της περιοχής. Αν υπάρξει αυτή τη στιγμή μια συμφωνία ελευθέρω εμπορίου με το Βιετνάμ, ε, όλη η περιοχή θα δει ότι θα υπάρχουν συνέπειες για την παραγωγή τους, για όλες τις παραγωγήσεις που θα μπορούσαν να γίνουν ε, στα πλαίσια της συμφωνίας με το Βιετνάμ, διότι το Βιετνάμ Α, συγγνώμη, είπα το Βιετνάμ, αλλά είναι η Ταϊλάνδη. Η Ταϊλάνδη είναι η πιο ανταγωνιστική χώρα όσον αφορά την ε, παραγωγή κονσέρβας τόνου. Η Παππούα Νέου Γουινέα έχει 0% δασμού στην ε, παραγωγή κονσερβοποίησης, αλλά ε, και η Ταϊλάνδη έχει 20%, αλλά αυτή είναι μια διαφορά που θα μπορούσε να είναι πολύ σημαντική. Τι εννοώ. Πρόκειται για μια αγορά που έχει πάρα πολλέ συνέπειε ε, ανάλογα με τι συμφωνίε που κάνουμε και εμεί. Και αυτό σα το λέω στα πλαίσια και μια στρατηγική η οποία θα πρέπει να είναι και εμπορική στι μελέτε που κάνουμε. Σας είπα προηγουμένως ότι παρά το γεγονός ότι ο ειρηνικός είναι πολύ μεγαλύτερος ε, εγώ θα σταθώ σε μερικά σημεία και για μας είναι πολύ πιο σημαντικό να σταθούμε στο κεντρικό και δυτικό ε, ειρηνικό κενό. Γιατί εκεί έχουμε τη μεγαλύτερη παραγωγή. Όπως σας είπα, ε, έχουμε το 80% της παγκόσμιας παραγωγής ε, του τόνου. Το 60% είναι στο κεντρικό και δυτικό ειρηνικό κενό. Και στην έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μετά θα πούμε και τι κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει ένα πρόβλημα ε, και άναρχης αλίας, παράνομης λαθρέας και άναρχης αλίας ε, στην περιοχή αυτή, διότι είναι 15 χώρες ακέ της περιοχής του Ειρηνικού εκεί, που η κάθε μία ενδιαφέρεται και για τη στρατηγική που θα κάνουμε στο μέλλον, και επιπλέον ε, γιατί η στρατηγική της ε, Συμφωνίας ε, Οικονομικής ε, Εταιρικής Σχέσης έχει σημασία για την περιοχή. Οι χώρες ΑΚΕ, όπως γνωρίζετε, ομαδοποιούνται σε 7 κατηγορίες. Έχουμε ειρηνικό, καραϊβική και εμάς μας ενδιαφέρει κυρίως αυτή η περιοχή του ειρηνικού δεν θα σας πω λεπτομέρειες, έχουμε τα νησιά Κουκ, ε, τη Μικρονησία, το Τουβάλου, τα νησιά του Σολομόντα. Είναι γνωστές λοιπόν οι 15 χώρες, δεν θα, σας τις πω με τη σειρά τις, έχουμε την Παππού Νέα και ούτε καθεξής. Οι χώρες αυτές είναι όλες μέλη της Περιφερειακής Οργάνωσης ε, του Δυτικού και Κεντρικού Ειρηνικού και με αυτές έχουμε συμφωνίες. Οι χώρες αυτές λοιπόν που έχουν την ιδιαιτερότητα να είναι χώρες ε, νήσι που είναι και το βασικό τους χαρακτηριστικό όλοι όσοι είμαστε από τα νησιά η συνάδελφος εδώ είναι από τις ε, Αζόρες ε, γνωρίζει γιατί μιλάω ο κύριος πρόεδρος ο οποίος επίσης προέρχεται από μια υπερπόντια περιοχή Πρόκειται για χώρες λοιπόν οι οποίες έχουν κάποιες ιδιαιτερότητες που δεν έχουν οι χώρες στις οποίες ζούμε εμείς στην υπηρετική Ευρώπη. Και πρέπει να πούμε ότι έχουν μία παραδοσιακή σχέση περιφερειακής διασύνδεσης σε όλους τους τομείς. Εγώ θα επικεντρωθώ βέβαια στον τομέα της αλίας και, και εκεί υπάρχει μια παραδοσιακή περιφερειακή σχέση και υπάρχουν ε, δύο περιφερειακές οργανώσεις που είναι πολύ σημαντικές. Η μία από αυτές είναι το Φόρουμ των Νησιών του Ειρηνικού, από το οποίο εξαρτάται και το Φόρουμ για την Αλία, FFA και υπάρχει το τμήμα της συμφωνίας του Ναούρου ε, PNA. Έτσι είναι γνωστό και έτσι θα το αναφέρω για να μην σας λέω όλα τα αρχικά. Από την άλλη πλευρά τώρα, του έχουμε και όλες αυτές τις τρίτες χώρες και εδώ βλέπουμε ε, πόσο ασχολούνται σε περιφερειακό από αυτά ε, επίπεδο οι χώρες αυτές. Έχουν συμφωνίες με τη ΣΥΠΑ από το 1988 και μάλιστα έχουν υπογράψει συμφωνία με την FFA που είναι η ε, το αλληλευτικό φόρουμ αυτού του φόρουμ συνεργασίας υπογράφει για το 2003 έως το 2013 και τώρα είμαστε στη διαδικασία της νέας διαπραγμάτευσης. Αυτή τη στιγμή η συμφωνία δίνει δυνατότητα πρόσβασης στις ζώνες αλίευσης αυτών των χωρών σε 55 αλλιευτικά σκάφη των Ηνωμένων Πολιτειών για ένα ποσό της τάξης των 14 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως. θα υπάρξει η νέα διαπραγμάτευση. Έχω απλώς κάποια προσεγγιστικά στοιχεία. Δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα οι διαπραγματεύσεις ε, για τη συμφωνία αυτή, αλλά αυτά τα οποία διαθέτω εγώ λένε ότι στη μελλοντική συμφωνία ε, σας είπα ότι τώρα έχουμε 55 και τώρα γίνεται διαπραγμάτευση μεταξύ 40 και 45. Θα μειωθεί ο στόλος κατά 10 ή 15 σκάφη για 8.000 ημέρες ε, αλίευσης, γιατί αυτό ήταν ε, τμήμα του συγκεκριμένου προγράμματος ε, ημερών αλίευσης που θα σας εξηγήσω αργότερα και είναι της τάξης των 60 εκατομμυρίων δολαρίων. είναι περίπου 6.000 δολάρια την ημέρα. Αν κάνετε και το λογαριασμό, περίπου βγάζουμε αυτό το ποσό. Και τώρα να περάσουμε στις διαπραγματεύσεις για την ε, Συμφωνία Οικονομικής Εταιρικής Σχέσης. Αυτή η συμφωνία, το λέω σε περίπτωση που δεν το γνωρίζετε, σημαίνει ότι θα ασχοληθούμε εκ νέου ε, με τις εμπορικές σχέσεις για τις χώρες και με την Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο να προσαρμόσουμε το σύστημα των γενικευμένων προτιμήσεων που προβλέπεται στη Συμφωνία του Κοτονού στις οδηγίες ε, και τις κατευθυντήρες γραμμές του ΠΟΕ, ε, ο οποίος αποφάσισε ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το σύστημα κατά αυτόν τον τρόπο, διότι αντιβαίνει στους κανόνες του ΠΟΕ και αυτό είναι ο νέος μηχανισμός ο οποίος προσπαθεί να ε, χρησιμοποιήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να ανανεώσει τη συμφωνία. Στην περιοχή του Ειρηνικού έγινε μια νέα διαπραγμάτευση για μια συμφωνία και είναι στη διαδικασία κύρωση διότι εμείς γνωμοδοτήσαμε και για αυτή τη συμφωνία ε, από πλευράς Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τον Ιανουάριο του 2011 κατόπιν το Συμβούλιο ενέκρινε τη συμφωνία το Φεβρουάριο και υπεγράφει από το Κοινοβούλιο της Παππούας Νέας Γουινέας τον Ιανουάριο ε, του 2013 και τα Φίτζι είχαν ε, πει ότι θα προσυπρογράψουν και αυτή τη συμφωνία, αλλά από ό,τι γνωρίζω προς το παρόν δεν την εφαρμόζουν. Σε αυτή τη συμφωνία λοιπόν εταιρική σχέση καθορίζονται σαφώς ε, ποιοι είναι οι στόχοι και οι στόχοι είναι να βελτιωθεί η πρόσβαση στην αγορά και να υπάρχει μια βιώσιμη ανάπτυξη και να υποστηρίζεται μια περιοχή ελευθέρου εμπορίου. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι για πρώτη φορά υπάρχει μια παρέκκληση, όπως θα θυμάστε, όλοι όσοι ήσασταν εδώ, των κοινοτικών κανόνων. Και αυτό έχει σημασία παρά το γεγονός ότι ακόμα ε, δεν είναι άξιες λόγου οι συνέπειες. Αυτός ήταν ο χρυσός κανόνες ε, στις ε, δασμολογικές παραχωρήσεις που κάναμε προς τρίτες χώρες όταν υπήρχε προτιμησιακό καθεστώς σε δασμολογικά ζητήματα. Τα προϊόντα στα οποία θα δίνονταν αυτή η δασμολογική προτίμηση θα έπρεπε να προέρχονται από τη χώρα δικαιούχο του προτιμησιακού καθεστώτος, απλώς και μόνον για να προστατεύεται η παραγωγή αυτών των χωρών. Αυτός ήταν ο χρυσός κανόνας που πάντα είχε αποτέλεσμα. Για πρώτη φορά όμως ε, ε, αν και νομίζω ότι πρώτη φορά ήταν σε άλλη χώρα, για πρώτη φορά να γνωρίζετε επισήμως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είναι στην περίπτωση αυτής της συμφωνίας ε, η παρέκκληση. Εδώ είχαμε τις διαφωνίες μας, ε, η κυρία Λεβίν θα το θυμάται, διότι εμείς εδώ θεωρούμε, τουλάχιστον η γνωμοδότηση που εγκρίναμε αυτό έλεγε, ότι η Γενική Διεύθυνση Trade δεν είχε αναλύσει επαρκώς τις συνέπειες που θα μπορούσαν να έχουν ε, τα μέτρα αυτά των κανόνων ε, προέλευσης για τον τομέα των μεταποιημένων προϊόντων και όχι τόσο από πλευράς Ευρωπαϊκής Ένωση, του οποίους επικρίναμε και αυτού ότι δεν έκαναν επαρκή ανάλυση, αλλά κυρίως για τις τρίτε χώρες, όπως σας εξήγησα προηγουμένως για τα μεταποιημένα προϊόντα, διότι οι χώρες και τι Αφρικέ ε, και οι χώρες ε, που βρίσκονται στην, ε, πιο κοντά στη Λατινική Αμερική και είχαν σημαντικέ δασμολογικέ προτιμήσει, θεώρησαν ότι ε, θα μπορούσε να τους επηρεάσει αρνητικά αυτή η παρέκκληση. Δεν θα υπεκταθώ περαιτέρω γιατί το συζητήσαμε τότε και η Επιτροπή γνωμοδότησε από αυτού η Γενική Διεύθυνση Trade, ε, και σας το λέω ειλικρινά γιατί τότε ήμουν πολύ επικριτική με τη Γενική Διεύθυνση Trade, έλεγα ότι δεν έκαναν τίποτα για τα λιευτικά θέματα και λοιπά, χωρίς να λάβουν υπόψη όλες αυτές τις αποχρώσεις που εξήγησα προηγουμένως για το πώς γίνεται το εμπόριο στην αγορά του τόνου. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πω ότι είναι πολύ ενδιαφέρουσα η σχέση. Δεν ξέρω αν πριν ε, ε λήφθησαν ε, σοβαρά υπόψη οι κριτικές μου, αλλά τουλάχιστον αυτή τη στιγμή έχει συνειδητοποιήσει η Γενική Διεύθυνση Trade ότι αυτό το θέμα δεν είναι κοινότυπο και κυρίως δεν είναι κοινότυπο επειδή μπορεί να έχει συνέπειες για άλλες χώρες και επιμένω για άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Γενική Διεύθυνση Trade αυτή τη στιγμή διαπραγματεύεται μια συμφωνία που θα αντικαταστήσει αυτή την ε, διάμεση συμφωνία στην οποία αναφέρθηκα και θα αφορά όλες τις χώρες και της περιοχής και όχι μόνο την ε, Παππούα Νέα και τα Φίτζη και δεν θα περιλαμβάνει μόνο εμπόριο αγαθών αλλά και υπηρεσιών. Αυτό είναι πολύ γενικό βέβαια. Ε, ήθελα να σας, δεν χρειάζεται να σας πω εδώ περαιτέρω τι κάνει η Γενική Διεύθυνση 3, αλλά για την αλληλεία να σας πω τι μου είπαν εμένα. Ε, ήταν πολύ επίμαχη στις διαπραγματεύσεις. Αυτό το κομμάτι ήταν επίμαχο. Γιατί οι συγκεκριμένες χώρες ζητούν μια συνολική παρέκκληση των κανόνων προέλευσης. Όχι μόνο για τα μεταποιημένα που ήδη για αυτές τις δύο χώρες είχε δοθεί, αλλά μια παρέκκληση που θα περιλαμβάνει και τα κατευσυγμένα και τα νομπα προϊόντα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την πλευρά της Ναι, πρόεδρε, διακόπτει ο πρόεδρος στην ομιλητρία. Ε, μια φορά σα μιλάω για αυτό το θέμα, δεν θα τα ξαναπώ. Μιλάτε 25 λεπτά, σα ε, το υπενθυμίζω απλώς. Ε, δεν έχουμε τίποτα άλλο σήμερα το πρωί. Ε, πώς δεν έχουμε, λέει ο πρόεδρος. Έχουμε και παραέχουμε. Μέχρι τι 12 μεσάνυχτα δουλεύαμε χτε το βράδυ. Εγώ βγήκα από εδώ τα μεσάνυχτα με την κυρία Ρόντουστ, έτσι. Το μόνο που σας λέω είναι ότι θα, την επόμενη φορά δεν σας τα ξαναπώ. Σας τα λέω για να τα ακούσει η Κομισιόν. Αν θέλετε το βουλώνω, ε. Όχι, όχι, να μην το βουλώσετε κυρία Φράγα. Απλά σας είπα να τελειώσετε. Ε, ε, έχω ακόμα αρκετά να πω. Γι' αυτό σας το λέω. Ε, εγώ ή δουλεύω σε βάθος ή δεν δουλεύω καθόλου. Είμαι ε, τελειομανής. Το έχω στο αίμα μου. Λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, φαντάζομαι ότι σας ενδιαφέρουν αυτά που σας λέω. Αν δεν σας ενδιαφέρουν, να σταματήσω. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζήτησε να ληφθεί υπόψη ω ενδεχόμενο αντιστάθμισμα σε αυτή την ε, πλήρη παρέκκληση ε, επί των κανόνων προέλευσης. Ζήτησε λοιπόν να ληφθεί υπόψη ε, η πρόσβαση στους αλευτικούς πόρους τις ε, αποκλειστικές οικονομικές ε, ζώνες αυτών των χωρών. Και όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 της Προσωρινής Συμφωνίας, μια καλή διακυβέρνηση του τομέα της Αλίας και μια βιώσιμη ανάπτυξη του ελευτικού τομέα αυτό με έμεση αναφορά στην παράνομη λαθρέα και αναρχιαλία κλπ. Συνεπώς ε, η συνολική παρέκκληση ε, να δοθεί, ζητάει η DigiTrade, ε, με αντιστάθμισμα πρόσβαση στην οικονομική τους, στην οικονομική τους ζώνη, στους αληθικούς πόρους αυτής της ζώνης και μια καλή διακυβέρνηση στο τομέα της αλίας. Προς το παρόν δεν, προέκυψαν, προέκυψε πρόοδος, οι διαπραγματεύσει έχουν μπλοκαριστεί, ο καθένας ζητάει το δικό του. Αλλά πιστεύω από τις πληροφορίες που έχω πάρει, οι χώρες ΑΚΕ δεν είναι πρόθυμες να αναζητήσουν μια λύση αυτή τη στιγμή. Πάντως, ένας επόμενος γύρος διαπραγματεύσεων θα ξεκινήσει τον Ιούνιο στις Βρυξέλλες. Γι' αυτό το λόγο ήθελα να καθυστερήσουμε λίγο τη συζήτηση για να δούμε τι θα γίνει αν ξεμπλοκαριστεί το θέμα. Τώρα, να κάνω κάποιες σκέψεις, προσωπικές σκέψεις, δικές μου, έχοντας αναλύσει την κατάσταση. Πρόεδρε, μη με κοιτάτε έτσι γιατί με κάνετε να γελάω. Σκέψεις μου λοιπόν. Αυτές οι χώρες ε, δίδουν, αποδίδουν τρομακτική σημασία στην Αλία. Αυτό πρέπει να το υπογραμμίσουμε. Θέλουν να διευρύνουν τις ε, παρεκκλήσεις των κανόνων προέλευσης, είναι προφανές αυτό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση από την άλλη μεριά δεν θέλει να διευρύνει αυτό το πεδίο χωρίς ε, κάποιο αντιστάθμισμα και σε πρόσβαση ελευθερικού πόρου, πόρους αλλά και σε από διακυβέρνησης, διαχείρισης του Μετσαλίας. Τώρα, δεν καταλαβαίνω πολύ καλά γιατί υπάρχει αυτό το ενδιαφέρον από την πλευρά αυτών των χωρών δεδομένων των δυσκολιών που έχουν εξαιτία υψηλού κόστους παραγωγής ε, και από απομακρυσμένη θέση τους σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, γιατί στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν μια ανταγωνιστική θέση εξαιτία αυτών των ε, μειονεκτημάτων που έχουν. Ε, για παράδειγμα με την Ταϊλάνδη. Η Ταϊλάνδη είναι πολύ πιο ανταγωνιστική στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε η μόνη εξήγηση που μπορώ να δώσω εγώ για το ενδιαφέρον που δείχνουν αυτές οι χώρες είναι ότι προσπαθούν να αυτοπροστατευτούν από τον κανονισμό για την παράνομη λαθρέα και αναρχιαλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα τώρα που ορισμένες από αυτές τις χώρες, Φίτζι και Βανουάτο, ε, που ε, έχουν ήδη ειδοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ άλλες χώρες ε, βρίσκονται υπό έρευνα, αποτελούν αντικείμενο έρευνας. Θα πρέπει να δούμε πώς θα ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις πάντως για να καταλάβουμε. Να δούμε αν πράγματι είναι δυνατή μια συμφωνία με κάποιο αντιστάθμισμα για μας ε, που θα μας ε, δίνει ενδεχομένως μια πρόσβαση στα υδατά τους. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια αύξηση της αλληλευτικής προσπάθειας. Σημαίνει απλώς ε, βελτίωση της πρόσβασης. Όλα αυτά θα πρέπει να τα διαχειριστούμε στο πλαίσιο ενός, σε ένα νομικό πλαίσιο το οποίο θα διαπραγματευτούμε ενδεχομένως και με την FFA. Ε, θα πρέπει να δούμε αν κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει σε συνεργασία και με την Κομισιόν ε, και όπως ε, είπα με την FFA θα πρέπει να δούμε πώς θα εφαρμοστεί μια τέτοια συμφωνία. Δεύτερον, ε, πώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν αυτά αργότερα μέσω διμερών συμφωνιών και ποιες θα πρέπει να είναι διατάξεις περί ε, διακυβέρνησης, διαφάνειας, καταπολέμησης τη και αναρχισαλίας κλπ. Η κυρία Λαβέν δεν με ακούει αυτή βέβαια, αλλά θα μπορούσε να με βοηθήσει γι' αυτό. για το σύστημα Best Day ε, βέλτιστης μέρας. Ε, θα μπορούσε να εφαρμοστεί ενδεχομένως υπό την προϋπόθεση ότι θα ε, ε σωστά και θα ήταν διαφανές. Εν πάση περιπτώσει, το πλαίσιο αυτό θα έπρεπε να είναι περιφερειακό θα συνοδεύεται από διμερείς συμφωνίες δηλαδή, αλλά αυτό το σύστημα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να περιλαμβάνει διατάξει για την καταπολέμηση παράνομης λαθρές και αναξιαλίας, ενδεχομένως και ένα σύστημα best day ε, για το μέλλον. Έχετε δύο πίνακες για αυτό το σύστημα best day, από όπου φαίνεται ότι το σύστημα αυτή τη στιγμή δεν είναι διαφανές, αν λειτουργεί σωστά θα μπορούσε να είναι θετικό, θα ήθελα να το συζητήσουμε, αλλά ενδεχομένω όχι σήμερα. Οπότε εδώ τελειώνω. Ευχαριστώ. Πρόεδρο. Ναι, θα ξαναπάρετε το λόγο, κύριε φράγκα, Μην ανησυχείτε. Να σα ακούσουμε την Κομισιόν αυτή τώρα. Sí, prefieren eh, primero intervenir los diputados, ε, Συνήθως ε, δίνουμε το λόγο στην Κομισιόν μετά τον εισηγητή, την εισηγήτρια και μετά παίρνουν το λόγο οι ευρωβουλευτές. Αλλά αν θέλετε να περιμένετε, όπως θέλετε. Να ακούσουμε τους ευρωβουλευτές πρώτα. Ωραία, και μετά ο λόγος στην Κομισιόν. Uh, Πρόεδρε, Μία σύντομη δήλωση θέλω να κάνω στο όνομα της κυρίας Μάισνερ που δυστυχώς δεν μπορεί να είναι παρούσα σήμερα. Αλλά θα ήθελε να τονίσει κάποιες τυχές της, αλίας, ε, της παράνομης λαθρείας και της αλίας ε, στην περιοχή. Πιστεύει ότι ένα συμβιβασμός ε, στην αλλιευτική στρατηγική θα εμβαθύνει τις σχέσεις των χωρών αυτών με την Ένωση και επίσης τονίζει ότι οι συμφωνίες, οι αλευτικές συμφωνίες εταιρικής σχέσης θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη <clears throat> την περιφερειακή συνεργασία ε, μεταξύ των χωρών αυτών ε, και θα πρέπει να αυξήσουμε την πολιτική συνοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή θα ε, πρέπει να θαρρύνει τις χώρες αυτές να συνεργάζονται μεταξύ τους. Ε, θα πρέπει να υπάρχει ολοκληρωμένη στρατηγική αλλιευτική στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σχετικά με τον τρόπο αλληλείας στην περιοχή και θα πρέπει να στοχεύσουμε στο πρόβλημα της παράνομης λαθρείας και άναρχης αλληλείας. Η κυρία Μάισνερ προσβλέπει στη στενή συνεργασία με την εισηγήτρια για την ανάπτυξη του θέματος αυτού στις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Λεβίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ Κάρμεν. Άκουσα πολύ προσεκτικά τις εξηγήσεις σου και δεν νομίζω ότι μακρηγόρησες διότι νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα το θέμα αυτό. Σε, συγχαίρω λοιπόν για την πρωτοβουλία που πήρε για την έκθεση αυτή. Νομίζω ότι είναι επίκαιρη και οι διαπραγματεύσεις ε, της νέας αριευτική ε, συμφωνίας εταιρικής σχέση με τις ε, χώρες του Ειρηνικού συνεχίζεται, έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό και είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ασχοληθούμε στην Επιτροπή Αλληλείας διότι προφανώς ο βασικός ε, φυσικός πόρος στην περιοχή είναι η αλληλεία και ακριβώς ε, με αυτό ασχολείται η Ευρωπαϊκή Ένωση όταν διαπραγματεύεται τη νέα συμφωνία ε, εταιρικής σχέσης με την περιφέρεια αυτή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να διατηρεί περιφερειακή προσέγγιση και θα πρέπει να έχουμε συνεπή, συνεκτική θέση, να έχουμε δηλαδή την ίδια προσέγγιση στις ε, ε, αλληλευτικές ε, συμφωνίες εταιρική σχέσης με την Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Να μην προσπαθούμε να δημιουργήσουμε διαφορές ανάμεσα στις χώρες, ούτε να παρέμβουμε στον τρόπο που οργανώνονται μεταξύ τους. Χάρηκα λοιπόν που η κυρία Φράγα τόνισε την συμφωνία του Ναουρού και τους διεθνείς οργανισμούς που ε, λειτουργούν εδώ και πολύ καιρό ε, στην περιοχή αυτή. Πρόκειται για ε, λιγότερο αμφιγμένες χώρες οι περισσότερες από αυτές τις χώρες και μάλιστα έχουν καταφέρει πολύ καλά να έχουν κοινή προσέγγιση για την υπεράσπιση των φυσικών του σπόρων, ιδιαίτερα των ηχθείων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα πρέπει να έχει συνεκτική θέση και όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις ε, για τις ελληνικές συμφωνίες εταιρική σχέσης. Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει καταφέρει να οριστικοποιήσει την ε, αλληλευτική συμφωνία με τη Μικρονησία ή της νήσου Σολομώντα, διότι υπήρχαν αρκετές εντάσεις ε, σχετικά με το μη σεβασμό της περιφερειακής προσέγγισης. και Γι' αυτό ε, έχουν ε, αποτύχει ε, αλλεπάλληλες συμφωνίες τέτοιες σχέσεις και με το να συναντούμε το ίδιο πρόβλημα, ότι η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης δημιουργεί σημαντικές εντάσεις στην περιοχή. Το Κυριμπάτι έχει υπογράψει συμφωνία χωρίς ε, μέρες ε, αλληλείας. Ε, του να αναφέρεται στην χωρητικότητα των πλοίων και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα τι αναπτυξιακέ πολιτικέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση, την εμπορική πολιτική τη Ευρωπαϊκή Ένωση και να έχουμε μια ολοκληρωμένη και συνεκτική πολιτική, μια ολοκληρωμένη και συνεκτική προσέγγιση προ τον έξω κόσμο. Δεν βοηθάει λοιπόν το γεγονός ότι στις ε, περιφερειακές οργανώσεις ε, αλληλείας ε, της περιοχής η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εικόνα μιας λιγότερο συνεργάσιμης οντότητας όσον αφορά την αλληλεία από την ανάπτυξη. Νομίζω ότι αυτό που τόνισε η κυρία Φράγα ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει πρόσβαση στους πόρους ε, στο πλαίσιο αυτή της ε, αλλιευτικής ε, συμφωνία εταιρική σχέσης. Οι πράσινοι δεν, δεν στηρίζουμε μια τέτοια προσέγγιση. Πιστεύουμε ότι οι πόροι των χωρών αυτών είναι δικοί τους, ανήκουν στις χώρες αυτές και ότι θα πρέπει να είναι δικαίωμά τους να αποφασίσουν σχετικά με τους πόρους αυτούς. Ξέρω ότι είναι πολύ ευαίσθητο το θέμα αυτό. Είδα το ποσοστό του 5% για το σύνολο των πόρων που θα πρέπει να είναι το όριο για την υπογραφή μιας ε, αληφτικής συμφωνίας εταιρικής σχέσης. Θα ήθελα να ρωτήσω την ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή αν ισχύει αυτό. Και όσον αφορά αυτό που Ζητάνε οι χώρες ΑΚΕ την, ε, ε, ε, την επέκταση της παρέκκλησης. Θα ήθελα να ρωτήσω την Κομισιόν τι γνώμη έχει γι' αυτό, τι συνέπειες θα έχει μια τέτοια παρέκκληση. Η Πατράου Νέβες. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, τις μου και στην Κάρμεν για την λεπτομερή παρουσίαση ενός τόσο περίπλοκου ζητήματος. Πολύ σημαντικού όμως που έχει μεγάλο αντίκτυπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό το ζήτημα. Θα είναι πολύ σύντομη ε, στην παρουσίαση των δικών μου ανησυχιών, ε, κυρίως επειδή μερικές από αυτές, πολλές από αυτές έχουν επανειλημμένως εκφραστεί και από μένα και από άλλους συναδέλφους εδώ. Αξίζει τον κόπο όμως να υπογραμμίσουμε κάποιες από αυτές τις ανησυχίες μία ακόμα φορά γιατί έχουν άμεση σχέση με αυτό που συζητούμε. Καταρχήν με ανησυχεί η ανακοίνωση Συμφωνίας Ελευθερών συναλλαγούμενη με την Ταϊλάνδη γιατί κάτι τέτοιο μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην, στο δικό μας κλάδο κονσερβοποίησης μεταποίησης. Αυτή τη στιγμή η Ταϊλάνδη ε, ε, ήδη εξάγει μεγάλο αριθμό κονσερβών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ορισμένες από τις ε, εξαγωγές της Ταϊλάνδης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, έχουν μειώθηκαν λίγο το 2012 ακριβώς διότι οι συνθήκες ε, ε παραγωγής των κονσερβών δεν ήταν επαρκής. Συνεπώς η, δεν διασφαλιζόταν η ποιότητα του προϊόντος. Γιατί, Γιατί οι απαιτήσει προς τους δικούς μας παραγωγούς δεν γίνονται σεβαστές πολύ συχνά από παραγωγούς τρίτων χωρών που εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι επίσης σαφές ότι ή οι κονσέρβες τόνου θα μείνουν εκτός της συμφωνίας ελεύθερων συναλλαγών με την Ταϊλάνδη ή ως ευαίσθητο προϊόν θα πρέπει να υπόκεινται σε ιδιαίτερη συγκεκριμένη και επαρκή προστασία. Γιατί περνάμε μια περίοδο κρίση στην Ευρώπη, δεν έχουμε την πολυτέλεια λοιπόν να ε, πνίξουμε ακόμα περισσότερο ε, έναν κλάδο, όχι μόνο βιομηχανικό, αλλά κυρίως το βιομηχανικό, που λειτουργεί παραδοσιακά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και από τον οποίο κλάδο εξαρτώνται πολλές θέσεις εργασίας Και μια οικονομική δυναμική πολλών χωρών του Νότου. Δεύτερο θέμα έχει σχέση με την ηχθειοκαλλιέργεια. Η ηχθειοκαλλιέργεια για την επόμενη μεταρρύθμιση της ε, κοινή αλληλευτικής πολιτικής θα είναι ένα μεγάλο στίχημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κατακλείζεται συστηματικά από προϊόντα ηχθειοκαλλιέργειας πρόλευσης Ασίας. Και πάλι με συνθήκες παραγωγής και μεταποίησης που είναι αντικείμενο πολλών επικρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλουμε να έχουμε διαφορετικούς κανόνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε τρίτες χώρες. Πολύ προσοχή λοιπόν, δεδομένου ότι ε, αναμένουμε μια σημαντική αύξηση της ε, ε της ηχθειοκαλλιέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τη μεταρρύθμιση που έρχεται. Τρίτον, θα πρέπει να είμαστε όλο και πιο αυστηροί σε ό,τι αφορά τις απαιτήσει ε, σεβασμού των ίδιων κανόνων εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι δυνατόν να ξεκινήσουν να μιλάμε ήδη για παρεκκλήσεις από τους κανόνες προέλευσης ή από άλλους κανόνες, δεδομένου ότι ε, επί τη βάση του νέου γράφου του ΠΟΕ γνωρίζουμε πως ε, οι υποχρεώσεις του ευρωπαϊκού τομέα, του, του, του κλάδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα γίνονται όλο και πιο αυστηρές. Έχουμε πάρα πολλά συμφέροντα ε, και η διαφορά ανάμεσα στους κανόνες που ισχύουν στην Ευρωπαϊκή, στους Ευρωπαίους παραγωγούς και στους παραγωγούς τρίτων χωρών, αυτή η διαφορά ε, μπορεί να αποβεί εις βάρος μας. Αυτά είναι τα τρία σημεία τα οποία ήθελα να υπογραμμίσω και θα ήθελα να ληφθούν υπόψη, ε, ενώ σε ό,τι αφορά τα πιο λεπτομερή θέματα θα τα δούμε στις επόμενες συζητήσεις μας. Ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια μια ακόμα φορά στην Κάρμεν για την εξαιρετική παρουσίαση που μας έκανε. Ευχαριστώ. Κυρία Τόμας. Oui, merci, Monsieur le Président. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την κυρία Φράγκα για την παρουσίαση αυτή. Πράγματι, όπω είπε και η ίδια, δεν είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία κατέχω εγώ καλύτερα, αλλά θα ήθελα, ε, θα ήθελα να θέσω ένα ερωτηματικό προς το παρόν. Καταρχάς, ε, θεωρώ ότι όπως είπε και η κυρία Λεβέ, είναι όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματεύεται μία ε, εμπορική συμφωνία με τις χώρες του ειρηνικού, προφανώς ένα μεγάλο τμήμα των συμφωνιών αυτών αφορούν την αλληλεία και αυτό διότι πρόκειται για ένα ε, φυσικό θαλάσσιο απόθεμα. Γι' αυτό λοιπόν θα πρέπει να εισακουστεί και η άποψη της Επιτροπής ε, σε αυτές τις διαπραγματεύσεις. Και επίσης θεωρώ ότι η στρατηγική αυτή και οι προϋποθέσεις αυτών των συμφωνιών ε, θέτουν την Ευρωπαϊκή Ένωση ενώπιον των ίδιων της των αντιθέσεων. Αφενός ε, έχουμε πολύ αυστηρές απαιτήσει ε, για την αντιμετώπιση της παράνομης αλληλείας ε, και της ε, λαθρέας και άναρχης, αλλά τουλάχιστον δύο χώρες, αν κατάλαβα καλά κυρία Φράγκα, οι οποίες είναι αντικείμενο έρευνας ή τουλάχιστον ελέγχου για παράνομη αλληλεία, έχουμε λοιπόν τουλάχιστον υποψίες για παράνομη αλία σε μια περίπτωση και ταυτόχρονα ου έχουμε συμφωνίες ε, με την Παππούα η Ινέα που λένε ότι δεν υπάρχει ε, παρέκκληση για τη χώρα προέλευσης. Επομένως, αν κατάλαβα καλά, για τα μεταποιημένα προϊόντα τη σήμερον ημέρα, αν δεν υπάρχουν κανόνες ε, για τη χώρα προέλευσης, θα μπορούσαμε να έχουμε προϊόντα τα οποία προέρχονται από χώρες που έχουν ως πρακτική τους την παράνομη Και ξαφνικά είμαστε διατεθειμένοι να γενικεύσουμε την κατάσταση. Θα χάσουμε λοιπόν οποιονδήποτε τρόπο ελέγχου και θα διευκολύνουμε ε, τις... Ε, ε, μεταφορές ε, παράνομων αλλιευμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πραγματικά μου δημιουργούνται ερωτηματικά, κυρία Φράγκα. Ποια είναι η καλή λύση. Η καλή λύση θα ήταν να μην δεχτούμε παρεκκλήσεις για τους ε, κανόνες της χώρας προέλευσης ή θα πρέπει να μην υπάρχουν δικαιώματα πρόσβασης σε ζώνες αποκλειστικής οικονομικής εκμετάλλευσης. Εγώ θεωρώ, έτσι ενθερμό, ότι θα έπρεπε να υπάρχουν κανόνες ώστε οι εμπορικές μας συμφωνίες να έχουν και περισσότερες απαιτήσει. Ε, και νομίζω ότι με αυτή τη γενίκευση των εξαιρέσεων ε, για τη χώρα προέλευσης ουσιαστικά ε, αφήνουμε το ελεύθερο για οποιαδήποτε παραβίαση των κανόνων, ε, απουσία πλήρη κανόνων, ακόμα και διευκόλυνση της παράνομης αλίας. Πραγματικά αυτό μου έρχεται εδώ ως ε, αντίδραση στην πρώτη συζήτηση. Ευχαριστώ κυρία Τόμας. Τώρα να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τον κύριο Πίπερ. Yes, uh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Σύμφωνο με τις προηγούμενες παρατηρήσεις. Είναι εξαιρετική η περιγραφή αυτή, πολύ καλή εισαγωγή στη συζήτηση και πολύ ευχαρίστως ε, θα σχολιάσω κάποια στοιχεία και θα απαντήσω και σε κάποιες ερωτήσεις. Καταρχήν είναι απόλυτα σωστό ότι η περιοχή αυτή παράγει το μεγαλύτερο μέρος του τόνου του κόσμου και θα πρέπει ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση να φερθεί υπεύθυνα και να προσεγγίσει από αυτή την άποψη το θέμα. Ε, το πλαίσιο είναι η συζήτηση για την ε, Συμφωνία Εταιρικής Σχέσης. Βρισκόμαστε σε, στενή συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση ε, Εμπορίου. Εξετάζουμε την πρόοδο που σημειώνεται. Εξετάζουμε και την πρόσβαση των χωρών του, ωκεανού, του Ειρηνικού ωκεανού στην ευρωπαϊκή αγορά. Έχουμε προσθέσει και στοιχεία ε, ε, διατήρηση του περιβάλλοντος ε, και καλή διακυβέρνησης. Είναι μία δήλωση προς τις αγορές και θέλουμε να φερθούμε υπεύθυνα. Παρότι πρόκειται για εμπορική συμφωνία προς όφελος του εταίρου μας, θα πρέπει να υπάρχει και όφελος για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να υπάρχει κάποια περιορισμένη πρόσβαση της, του στόλου μας ε, στους πόρους των νήσων αυτών. Όπως ανέφερε η κυρία Φράγα, έχουμε κάποια πρόσβαση στην περιοχή αυτή. Είναι πάρα πολύ περιορισμένη όμως. Ε, όσον αφορά το, τους γρήπους, το γρηγρή, ε, μιλάμε για τέσσερα σκάφη. <clears throat> Είναι λοιπόν πολύ περιορισμένη η πρόσβαση. Να αναφερθώ σε ένα από τα θέματα που αναφέρθηκαν. Ε, συνομιλούμε με τους συναδέλφους μας στη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Ναι, πράγματι. Και στο πλαίσιο αυτό σημαντικά στοιχεία της παρουσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή είναι ε, η παρουσία μας στις περιφερειακές οργανώσεις αλληλείας. Αυτό αναφέρθηκε πολύ σωστά. Και εδώ επιδιώκουμε να εργαζόμαστε με βάση την επιστήμη και προς ε, την ε, διατήρηση των αποθεμάτων. Ε, θέλουμε δηλαδή να καθορίζονται οι τιμές με βάση τι επιστημονικέ αξιολογήσει, κάτι που ευθυγραμμίζεται απόλυτα με αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Θέλουμε επίση συμμόρφωση με του κανόνε και καλή διακυβέρνηση. Έχουμε λοιπόν ε, ένα αυτόνομο εργαλείο για την καταπολέμηση της ε, παράνομης λαθρείας και αναρχής αλληλείας. Ε, ξέρετε ότι αυτό γενικά είναι ένα θέμα με το οποίο ασχολούμαστε. Έχουμε αναλύσει κάποιες από τις χώρες της περιοχής και μπορώ να σας πω ότι παρακολουθούμε το θέμα αυτό. Αναλαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα βήματα. Ξέρετε ότι πρέπει να υπάρχει διάλογος, να υπάρχει δυνατότητα σχολιασμού. Όλα αυτά πάνε πολύ καλά και υπάρχουν κάποιες χώρες της περιοχής ε, που συμμετέχουν στις εργασίες αυτές. Στα πλαίσια λοιπόν της Περιφερικής Οργάνωσης Αλληλείας ακολουθούμε τις κατευθυντήρες γραμμές ε, που παρεπτόντως έχει υποβάλει το κοινοβούλιο σας. Όσον αφορά τα στοιχεία της διμερούς συνεργασίας, έχουμε πάντα την ε, υπογραφή συμφωνιών εταιρικής σχέσης ε, και έχουμε τώρα συμφωνία με το κυριπάτι την οποία έχετε μπροστά σας και ελπίζω ότι θα μπορέσετε να συμφωνήσετε με την συμφωνία αυτή, ευθυγραμμίστε απόλυτα με τις κατευθυντήρες γραμμές που μας έχετε δώσει. Έχουμε αύξηση του ε, μεγέθους του στόλου, ε, έχουμε τομεακή συνεργασία, έχουμε αποσύνδεση των τελών πρόσβασης ε, και της τομεακής συνεργασίας, έχουμε ρήτρα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομίζω ότι όλα αυτά είναι σε μεγάλο βαθμό προς όφελος του, του Κυριμπάτη και συμφωνούν, συμφωνεί απόλυτα το Κυριμπάτη με τη συμφωνία αυτή. Στο πλαίσιο αυτό προέκυψε το θέμα τι κάνουμε με το πρόγραμμα ε, ημερών ανασκάφος, ημερών αλληλείας. Και η απάντηση είναι ότι δεν είμαστε κατά του προγράμματος αυτού του BDS. Μπορεί να είναι πολύ καλό, αλλά δυστυχώς ο τρόπος με τον οποίο ε, έχει διαμορφωθεί τώρα δεν είναι ικανοποιητικός και γι' αυτό δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να εγκρίνουμε το πρόγραμμα αυτό τη στιγμή που βλέπουμε ότι λείπουν ε, ε, σημαντικά μέρη, σημαντικά κομμάτια, όπως είναι για παράδειγμα η διαφάνεια. Θέλουμε να είναι πιο διαφανές, ε, να μην προκαλεί διακρίσεις, θέλουμε οι προϋποθέσεις να κοινοποιηθούν ώστε ο κόσμος να γνωρίζει πώς εφαρμόζεται το πρόγραμμα αυτό. να διασφαλίσουμε κιόλα ότι το πρόγραμμα αυτό συνάδει με τις επιστημονικές ε, συμβουλές, σε κάτι που δεν συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν είμαστε λοιπόν κατά του προγράμματος αυτού του καθεαυτού, το συζητάμε ε, με τις περιφερειακές οργανώσεις ε, στον Ειρηνικό. Πήγαμε εκεί και τους αντίσαμε, έχουν έρθει και εκείνοι εδώ ε, έχουμε συζητήσει λοιπόν το θέμα και γνωρίζουν πολύ καλά ότι είμαστε διατεθειμένοι να ε, ασχοληθούμε με το θέμα, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα το στόχο μας. Ε, στο μεταξύ ελπίζουμε ότι το θέμα του Κυριμπάτη μπορεί να προωθηθεί και να μας επιτρέψει να παραμείνουμε στην περιοχή και να συνεχίσουμε να παίζουμε ένα ρόλο στην περιοχή, έστω και ελάχιστο. Εμείς λοιπόν ως Ευρωπαϊκή Ένωση έχουμε πολύ περιορισμένη παρουσία εκεί και σίγουρα ε, δεν, διακινδυνεύει, δεν διακινδυνεύουν τα αποθέματα ε, ε, λόγω του δικού μας στόλου. Έχουμε συνάψει συμφωνία με τη Μικρονησία, δυστυχώς όμως... Να το θέσω ως εξής, εμείς σεβαστήκαμε όλα τα στοιχεία της συμφωνίας, αλλά η Μικρονησία δεν το έκανε, ήταν ατυχής η κατάσταση αυτή, γι' αυτό έπρεπε να αποσύρουμε το πρωτόκολλο αυτό σε συμφωνία με, το, με τη Μικρονησία και ε, οι νήσοι Σολομώντα έχουν κολλήσει. Ε, έχουμε προχωρήσει όμως ε, ως προς την εξέταση νέων συμφωνιών ε, με τις νήσους Κουκ. Προχωράμε και σύντομα θα υπάρξει η εντολή διαπραγματεύσεων και οι διμερείς επαφές προχωράνε πολύ καλά. Επίσης, τέθηκε ερώτηση, μπορούμε να έχουμε ολοκληρωμένη προσέγγιση όσον αφορά τις ε, ε, συμφωνίες εταιρικής σχέσης. Ε, ναι, ε, έχουμε και τεχνική προσέγγιση, αλλά σίγουρα μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο. Πολύ σημαντικό εδώ είναι όλα αυτά να γίνουν σε ένα πλαίσιο με προβλέψιμες συνθήκες εργασίας, να υπάρχει δηλαδή νομική βεβαιότητα. Να γνωρίζουμε πώς μπορεί να ε, κινηθεί ο στόλος, ε, όλα αυτά να ε, ε, βασίζονται σε επιστημονικές σύμβουλες και να είναι σαφείς οι στόχοι όσον αφορά τη διατήρηση των αποθεμάτων. Ε, ενώ δηλαδή στην περιφερειακή ε, οργάνωση αλίας υπήρχε ε, προσπάθεια μείωσης της αλίας, είδαμε ότι οι μέρες αλίας των σκαφών αυξάνονταν. Αυτή τη στιγμή λοιπόν συνομιλούμε με τους εταίρους μας. φροντίζουμε όμως να μην γίνουν διακρίσεις εις βάρος του αλευτικού μας τόλου. Όπως υπόθηκε, θα πρέπει να υπάρχουν ε, συνθήκες ίσου ανταγωνισμού. Και εφόσον έχουμε ήδη μικρή παρουσία ε, στην περιοχή, δεν μπορούμε να δεχτούμε ε, διακρίσεις εις βάρος των σκαφών μας. Επίσης, τέθηκε ερώτηση σχετικά με την πρόσβαση και ζητήθηκε ε, από την Ευρωπαϊκή Ένωση ποσοστό 5% πρόσβασης. Ε, όχι, το 5% αυτό παρεπιπτόντος προέκυψε από μια συζήτηση όπου αν θυμάμαι καλά η πλευρά του ελληνικού ρώτησε 5% και είπαμε εντάξει 5%. Αλλά το θέμα δεν είναι ότι θέλουμε 5% και το 4% δεν αρκεί. Το θέμα είναι να δημιουργήσουμε μια πλατφόρμα και να συζητήσουμε με ισορροπημένο τρόπο κάποιου είδους πρόσβαση για μας. Κατά τα άλλα όμως να διασφαλίζουμε ως ε, υπεύθυνο φορέας να έχουμε κάποιες διασφαλίσεις ε, σωστής διαχείρισης του συνόλου του συστήματος. Αυτή είναι σημαντική πτυχή και οι συζητήσεις συνεχίζονται. Επίσης, τέθηκαν ερωτήσεις σχετικά με το global sourcing. Τι συνέπειες έχει, τι σημαίνει. Είναι πολύ τεχνικό το θέμα αυτό. Μιλάμε για παρέκκληση στους ε, παραδοσιακούς κανόνες ε, προέλευσης ε, που υπάρχουν στις συμφωνίες ελεύθερου εμπορίου. Συνήθως γίνεται διμερώς σε μια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου. Δεν μιλάμε για μια παγκόσμια συμφωνία, μιλάμε για μια διμερή συμφωνία. Και αν έχουμε μια σειρά διμερών συμφωνιών, φροντίζουμε τα ωφέλη να ε, ε, ε, καθορίζονται στη συμφωνία αυτή. Έχουμε λοιπόν μια παρέκκληση σχετικά με το global sourcing και ποιες είναι οι συνέπειες να χάνουμε τον έλεγχο του, του, τι συμβαίνει. Ποιος είναι ο κίνδυνος. Ο, ο κίνδυνος είναι να έχουμε έναν στόλο παράνομης λαθρείας και αναρχής αλληλείας τον οποίο να μην μπορούμε να ελέγξουμε καθόλου και έτσι να μην μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Άλλος κίνδυνος ε, είναι ε, ο εταίρος μας να μην αποφελείται, ε, το μεγαλύτερο μέρος του κέρδους δηλαδή να πηγαίνει αλλού. σε κάποιον με τον οποίο ενδεχομένω επίση να διαπραγματευόμαστε. Λοιπόν, δεν είναι καλή ιδέα να ανοίγουμε παραθυράκια με τις παρεκκλήσεις αυτές για τρίτους που δεν ε, είναι συμβαλόμενα μέρη της Δημερού συμφωνίας. Αυτός είναι ο κίνδυνος και ο κίνδυνος λοιπόν είναι άλλοι ασιατικοί στόλοι να επωφεληθούν από αυτή τη ρήτρα. Και εμέσως να δοθεί πρόσβαση στην αγορά σε πολλούς ε, άλλους ξένους στόλους. Κάποιοι μέρος του όφελους ε, το λαμβάνει ο εταίρος μας, αλλά ε, αυτό είναι και θέμα κρίσης. Ε, μπορεί ουσιαστικά δηλαδή να χαρίζουμε κάτι σε άλλους, την πρόσβαση στην ευρωπαϊκή αγορά και το μεγαλύτερο μέρος του κέρδους να πηγαίνει σε κάποιον άλλον και όχι στο συμβαλόμενο μέρος. Το θέμα λοιπόν είναι υπάρχει αρκετό όφελος για ε, τη χώρα με την οποία συνομιλούμε ή πηγαίνουν αλλού τελικά τα κέρδη. Θα πρέπει αυτά να τα πολύ προσεκτικά. Θα πρέπει να δούμε λοιπόν μήπως έχουμε άλλα μέσα πιο κατάλληλα. Στο πλαίσιο αυτό θα πρέπει επίσης να φροντίσουμε ε, θα πρέπει να εξετάσουμε το όφελος. Ε, θα πρέπει να δούμε τελικά λοιπόν εάν το όφελος αυτό διαβρώνεται εντός εισαγωγικών, εάν υπάρχουν αρνητικές ε, συνέπειες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και εάν τελικά δεν έχουμε συνθήκες ίσου ανταγωνισμού, εάν δηλαδή εκχωρήσουμε κάτι, να φροντίσουμε να υπάρχει σωστή ισορροπία. Νομίζω ότι απάντησα λίγο πολύ στις περισσότερες ερωτήσεις και παρατηρήσεις. Και βέβαια είμαι στη διάθεσή σας ε, αν έχετε περισσότερες απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κυρία Φράγα. Η Κομισιόν απάντησε σχεδόν σε όλα, αλλά ήθελα να πω μερικά άλλα ακόμα πράγματα. Ε, η παγκόσμια ή περιφερειακή ε, συγκέντρωση. Ε, εγώ συμφωνώ με αυτό, θα πρέπει να εστιάσουμε σε παγκόσμιο και περιφερειακό επίπεδο. Τώρα για το Vessel Day Scheme. Είμαι υπέρ ενός τέτοιου συστήματος θα μπορούσε να γίνει δεκτό. Αλλά πρέπει να είναι διαφανές γιατί για να γίνει αυτός ο πίνακας όπου βλέπουμε ότι δεν συμμορφώνονται με το ε, Vessel Day Scheme χρειάστηκε να χρησιμοποιήσω τα τελευταία στοιχεία του WCPFC που διαφέρουν κατά 20% έως 20% με τα αρχικά στοιχεία που είχα εγώ. Για το 2009 η πόδα κεντρικού και δυτικού Ατλαντικού ε, Ελληνικού ωκεανού ε, ενέκρινε ένα όριο αλληλευτικής προσπάθειας που θα έπρεπε να είναι ο μέσος όρος των ετών 2002 με 2004 αν θυμάμαι καλά. Όμως δεν συμμορφώθηκαν με αυτό το όριο όπως το βλέπετε. Το Vessel Day Scheme μπορεί να λειτουργεί σωστά, μπορεί να είναι ένα σωστό σύστημα. Αλλά η αρχή του θα πρέπει να είναι η διαφάνεια και θα πρέπει να τηρούν τη στόχη του. Αυτό δεν έχει επιτευχθεί μέχρι τώρα. Τώρα, σε ό,τι φορά τα όσα είπε η κυρία Πατράου, συμφωνώ. Και δεν είναι μόνο ο αντίκτυπος που θα μπορούσε να, μπορούσαν να έχουν αυτά, αυτές τις προτάσεις σε εμά, αλλά και στις τρίτες χώρες. Νομίζω ότι αν υπογραφεί η Συμφωνία Ελεύθερης, ε, Ελεύθερης με την Ταϊλάνδη, με μηδενικούς δασμούς για τις εξαγωγές της Ταϊλάνδης, όλη η εμπορική πολιτική υπέρ των χωρών αυτών στον κλάδο της αλίας θα ναυαγήσει, θα ναυαγήσουν, θα ναυαγήσει αυτή η προσπάθεια. Η Αυστραλία εισάγει πολλές ε, κονσέρβες από την Ταϊλάνδη, παλιότερα από την Παππούα Νέα Γουινέα, τώρα πια είναι η Παππούα Νέα Γουινέα, δεν μπορεί να ανταγωνιστεί τους μηδενικούς δασμού τη ε, δασμούς της ε, Ταϊλάνδης, οπότε δεν μπορεί να εξάγει στην Αυστραλία. Το ίδιο θα γίνει και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε αυτό που προσπαθώ να πω είναι ότι και από αναπτυξιακή πλευρά, κάτω από το αναπτυξιακό πρέσμα, οι εμπορικέ μα πολιτικέ έχουν επίδραση στις χώρες αυτές και μπορεί να επηρεάσουν του, ή μπορεί να επηρεάσει τους στόχους μας. Τώρα, για την κυρία Τομάς. Πρόκειται για μια αλλιευτική ζώνη που χαρακτηριζόταν παραδοσιακά από παρανομία και λαθρέα άλλια. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχει μια συγκεκριμένη διαδικασία όταν ερευνούμε χώρες οι οποίες ε, δεν συμμορφώνουν τον κανόνα IUU με τον κανονισμό IUU. Ε, υπάρχουν δύο χώρες, η Βανουάτου και η Φίτζη, οι οποίες έχουν ήδη προειδοποιηθεί. Αυτή είναι η δεύτερη φάση. Η πρώτη φάση είναι της έρευνας και υπάρχουν χώρες οι οποίες ε, ήδη ερευνώνται. Άλλες χώρες αυτής της περιοχής. Τώρα, το global sourcing, οι κανόνες προέλευσης. Ό,τι είναι να γίνει έχει γίνει. Διότι μόνο η Παππούα Νέα Γουινέα έχει επαρκή υποδομή. Οι υπόλοιπε χώρε οι οποίε το ζητούν προσπαθούν να καταλάβω γιατί το ζητούν. Εγώ πιστεύω ότι θέλουν να προστατευτούν έναν του, του κανονισμού παράνομη άναρχη και λαθρέα αλεία. Δεν καταλαβαίνω, δεν βρίσκω άλλο λόγο. Πράγματι υπάρχουν τρίτες χώρες όπως η Ταϊλάνδη και οι Φιλιππίνες που πραγματικά επενδύουν και αλλιεύουν σε ε, οικονομικές, ε, πληθυντικές οικονομικές ζώνες της Νέα Νέας που δεν έχει αρκετά ζαλευτικά σκάφη, οπότε επιτρέπει στους άλλους να μπουν στα ύδατά τους. Το 40% του κόσμου παραγωγής είναι η πρώτη ύλη. Γιατί πρόκειται για ε, ζώνες, ε, αποκλειστικές ε, οικονομικές ζώνες πολύ πλούσιες σε φυσικούς πόρους, γι' αυτό λόγο και προσελκύουν και ζαλευτικά σκάφη από τρίτες χώρες. Αυτά βασικά. Η πρόσβαση στους αληφτικούς πόρους είναι σημαντική, γιατί παρόλο ότι δεν θα αυξηθεί ο αληφτικός μας τόλος, δεδομένων των μέτρων του Δυτικού Κεντρικού Ειρηνικού, έχουμε μόνο ε, τέσσερους, τέσσερα σκάφη με γρήπους. Αλλά η παρουσία μας είναι σημαντική γιατί εκεί πάνω από 80% είναι ύδατα που ανήκουν σε ΑΟΣ. Είναι ελάχιστο το ποσοστό που είναι διεθνή Πρόκειται για ε, νησιωτικά κράτη που έχουν μεγάλες οικονομικές ζώνες, οπότε είναι σημαντικό να διασφαλίσουμε έστω και για αυτά τα τέσσερα σκάφη μας πρόσβαση σε αυτές τις ΑΟΣ. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος που να θέλει το λόγο, να περάσουμε στο επόμενο σημείο, τροποποίηση του κατανονισμού για τη διατήρηση μέσω τεχνικών μέσων για τα λευτικά αποθέματα της ε, Βαλτικής θάλασσας, ε, των Μπέλτ και του Σούντ. Πρόκειται για έναν κανονισμό που θα μας παρουσιάσει καταρχάς ο εισηγητής, ο κύριος Γκρόμπατσικ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο στη διάθεσή μας. Η έκθεση αυτή έχει συζητηθεί αρκετές φορές στο παρελθόν. Ε, είχαμε και συνεδριάσεις μεταξύ των σκεδών ισορροπητών και του φαινομένου και έχει συζητηθεί και εδώ στην Επιτροπή μας. Συμφωνήσαμε ότι η διαδικασία που θα εφαρμοστεί θα είναι η συνήθις διαδικασία για την τροποποίηση τεχνικών μέτρων για την Βαλτική θάλασσα, τα Μπέλτ και το Σούντ και θα θέλαμε να εφαρμόσουμε τις αρχές της συνθήκης της Λισαβόνας εδώ. Αρκετές φορές είχε αναφερθεί ότι πρόκειται για μια σημαντική έκθεση για το μέλλον της αλίας και τη διατήρηση των διαφόρων αποθεμάτων, ιδίως στην Βαλτική. Ωστόσο, Υπάρχουν δύο εκθέσει, οι οποίες είναι υποδιαπραγμάτευση από αυτή τη στιγμή που έχουν επηρεάσει την ε, κατάσταση. Ε, ελπίζουμε λοιπόν να ολοκληρωθούν αυτές οι διαπραγματεύσεις ε, σύντομα και Επίσης μας ενδιαφέρει το Ταμείο Αλίας και τη τελική απόφαση για το Ταμείο Αλίας. σίγουρα θα επηρεάσει ιδιαίτερα το θέμα αυτό. η Ευρωπαϊκή Επιτροπή άλλαξε την ε, προθεσμία για την ε, υποβολή τροπολογιών και έχουμε καθυστερήσει ιδιαίτερα. Ε, μετά από ένα χρόνο θα τεθεί σε ισχύ μετά την επίσημη δημοσίευση στην εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χρειάζεται όμως αρκετός χρόνος για να μπορέσουμε να αποφασίσουμε ε, τι ακριβώς θα γίνει. Λαμβάνουμε αρκετές πληροφορίες από αλληλείς που αλλιεύουν στη Βαλτική θάλασσα. Προσφάτως ε, έγιναν και κάποιες ε, συναντήσεις με αλληλευτικές οργανώσεις, όχι μόνο σε μία χώρα, την Πολωνία από την οποία κατάγομαι φυσικά, αλλά και σε άλλες. Οι συνεδριάσεις αυτές έγιναν σε πολλές άλλες χώρες γύρω από τη Βαλτική θάλασσα και είναι πάρα πολύ σημαντικό να σας αναφέρω εδώ τα συμπεράσματα από αυτές τις συνεδριάσεις. Εγώ συμμετείχα σε μία από αυτές τις συνεδριάσεις, στην Ούστκα για την αλληλεία του γάδου και εκεί υπάρχει εξειδίκευση στη συγκεκριμένη περιοχή. Αλλιεύεται γάδος ε, πρωτίστως και αναφέρθηκε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Είναι πολύ χαμηλής ποιότητας ο γάδος που αλλιεύεται εκεί. Αυτή τη στιγμή τα αποθέματα ναι μεν είναι υψηλά, διότι καταφέραμε να έχουμε ανασύσταση του είδους, αλλά η ποιότητα είναι πραγματικά καταστρεπτική. Στις συγκεκριμένες συνεδρίες μας παρουσιάστηκαν και κάποια ψάρια και είδαμε ότι πραγματικά ε, φαίνεται ότι δεν υπάρχει αρκετή τροφή ε, για το γάδο, δεν υπάρχει κατάλληλη ισορροπία μεταξύ των ειδών ε, της Βαλτικής θάλασσας, έχει διαταραχθεί για κάποιο λόγο. Και αυτό επειδή ακριβώς και η Βαλτική είναι πολύ ιδιαίτερη θάλασσα, έχει συγκεκριμένες μονοκαλλιέργειες, δημιουργούνται προβλήματα. Οι αλληλείς μας είπαν ότι το γεγονός ότι σταμάτησε η μονοκαλλιέργεια και άρχισαν να αλλιεύονται και άλλα είδη συμπεριλαμβανομένων και πελαγικών ειδών ε, οδήγησε σε υποβάθμιση της ποιότητας του γάδου. Γι' αυτό λοιπόν και ξεπλάγησαν οι αλληλείς από την πρόσφατη απόφαση που δημοσιεύθηκε πέρσι, απόφαση την οποία έλαβε το Συμβούλιο, για την αύξηση των ποσοστώσεων για την αλληλεία πελαγικών ειδών στη Βαλτική και μείωση των ποσοστώσεων για το γάδο. Αυτό οδήγησε σε διαταραχή της ισορροπίας και αλλοί θεωρούν ότι αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ποιότητα του γάδου είναι τόσο χαμηλή. και θεωρούν ότι είναι τόσο χαμηλή που δεν μπορεί να απολυθεί όλας Πρέπει να απορρίπτονται τα αλλιεύματα, διότι ε, δεν είναι καλής ποιότητας και θα πρέπει να ε, να τονίσω εδώ ότι μας έδειξαν κάποια παραδείγματα. Πρόκειται για ψάρια τα οποία δεν έχουν σχεδόν καθόλου σάρκα. Είναι απλώς ε, λέπια και κόκαλα. Ε, αυτά δεν είναι ψάρια προς πώληση. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διότι τα τεχνικά μέσα είναι ε, πολύ σημαντικά. Τα τεχνικά μέτρα μεταφράζονται σε ποιότητα για τα αλλιεύματα. Και έχουν επίσης ε, θετικές ε, συνέπειες για τις υποδομές, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κοινή αλλιευτική πολιτική. Διότι αυτή είναι και η προσπάθεια που κάνουμε, να μειωθούν οι απορρίψεις. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μέλλον της Ευρωπαϊκής Αλίας και τη διατήρηση των αποθεμάτων να λαμβάνονται λοιπόν κατάλληλα μέτρα. Με βάση τις διαπραγματεύσεις μας αποφασίσαμε ότι προς το παρόν θα στηρίξουμε την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ακολουθήσουμε την συνήθη διαδικασία για την τροποποίηση του συγκεκριμένου κανονισμού, αλλά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις ε, οι οποίες ε, ε, σημαίνουν ότι το θέμα επίγει και θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στα συμπεράσματα του Συμβουλίου. Ευχαριστώ. Πριν δώσω το λόγο στην Κομισιόν, κυρία Λεβίν. Uh, ε, ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ τον εισηγητή για τη δουλειά του. Συμφωνούμε απόλυτα με την προσέγγιση της έκθεσής σας. Θα ήθελα να τονίσω αυτό που μόλις είπε ο κύριος Κροβάτσεκ σχετικά με την ποιότητα του γάδου ε, στην Βαλτική. Είναι κάτι που το ακούμε και από ε, Σουηδούς αλείς. Ε, είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει όχι μόνο με τη βιομάζα, με την ε, καλή διατήρηση του αποθέματος. Θα πρέπει να δούμε όμως ε, και το μέγεθος, την κατανομή στην ηλικία των ψαριών και την εξάπλωση του αποθέματος αυτού. Παλότερα λοιπόν είχαμε μεγάλα και μικρά ψάρια, ενώ τώρα ε, η γάδη είναι ε, ε, μήκους 35-38 εκατοστών, πολύ ισχνή και αυτό ανησυχεί τους αλληλείς. Παρότι λοιπόν τα νούμερα της ISIS φαίνονται τα στοιχεία της ISIS φαίνονται καλά, υπάρχουν ανησυχίες και υπάρχουν, στην... υπάρχουν ακόμα και αλληλείς στη Σουηδία που λένε ότι είναι υπερβολικά υπερβολικές υποσοστώσεις, ε, διότι θα πρέπει ε, να αποκατασταθεί το απόθεμα. Ήθελα λοιπόν, μια και το θίξατε, να δράξω την ευκαιρία να πω ότι ε, αυτή είναι και η δική μου εντύπωση και πρέπει να δούμε τη συνολική εικόνα όσον αφορά την αποκατάσταση των αποθεμάτων, να μην κοιτάμε μόνο να κοιτάμε και ε, το μέγεθος των ηχθείων ε, και την ε, κατανομή των ηλικιών εντός του αποθέματος. Η επόμενη ομιλητρία. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή, τον κύριο Κρόπατσα, και για την έκθεσή του. Η Κομισιόν μπορεί να στηρίξει τις τροπολογίες του αυτή τη στιγμή και Θα θέλαμε μια διευθύνση σχετικά με την τροπολογία. Ε, αυτό έχει να κάνει με τις ε, οδηγίες για τη ε, σύνταξη τροπολογιών για όλες τις ε, προτάσεις μας. Αναφέρονται οι εννέα μήνες πριν από την λήξη της εξουσιοδότησης. Χρειάζεται λοιπόν εδώ διευκρίνηση. Στο εννιάμινο αυτό η Επιτροπή δεν επιτρέπεται να προτείνει πράξεις κατ' εξουσιοδότηση. Πρέπει η έκθεση να υποβάλλεται ε, Εάν η έκθεση πρέπει να υποβάλλεται 9 μήνες πριν, θα πρέπει το σχέδιο να εκπονηθεί ε, τουλάχιστον 3 μήνες πρωτού υποβληθεί στο Κοινοβούλιο. Η παρέκκληση αυτή, λοιπόν, ισχύει για 1,5 χρόνο. Από νομικής ε, πλευράς, λοιπόν, χρειάζεται να διευκρινιστεί η τροπολογία αυτή για όλες τις ε, πράξεις. Όσον αφορά τις επιστημονικές συμβουλές για τη Βαλτική, οι συμβουλές της ISIS ε, θα υποβληθούν αύριο για την επόμενη χρονιά. Οι επιστήμονες συζητούν το συγκεκριμένο οικοσύστημα και τη διαχείριση των αποθεμάτων στη Βαλτική και πράγματι πρέπει να ληφθεί υπόψη η εξάπλωση των αποθεμάτων καθώς ε, και οι, οι, οι τιμές για τη βιομάζα. Η Βαλτική είναι ένα περιορισμένο οικοσύστημα ε, διότι δεν υπάρχει αρκετή τροφή στη θάλασσα για τα ψάρια και, και δεν είναι αλμυρή. Ε, θα ε, λοιπόν στη συνέχεια της συζήτηση για τα αποθέματα της Βαλτικής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριος Προβάτσικ. για την τροπολογία υπαριθμών 2. Πώς να σας το πω. Χρειάζεται περισσότερη διευκρίνηση. Και θα το κάνουμε αυτό κατά τη διάρκεια των διημερών μας συζητήσεων ε, και παρουσία των εκπροσώπων της νομικών υπηρεσιών. Η Κομισιόν σίγουρα χρειάζεται χρόνο να προετοιμάσει τη θέση της και να καταρτήσει ένα σχέδιο. Είμαστε ανοιχτοί. Θα το δουλέψουμε. Προκειμένου η έκθεση να είναι άριστη ε, και να δίνοντας τον χρόνο στην Κομισιό να κάνει καλά τη δουλειά της. Πρόεδρο, Πρόεδρος, ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης, σημείο 7. Συνέχεια πρέπει να στην εκχώρηση νομοθετικών αρμοδιοτήτων και στον έλεγχο των κρατών μελών τη άσκηση εκτελεστικών αρμοδιοτήτων τη Επιτροπή. Είχαμε ανταλλάξει απόψη για αυτό το θέμα. Α, σε σχέση με το προηγούμενο θέμα, τροπολογίε μπορούν να υποβληθούν μέχρι τι 5 Ιουνίου το μεσημέρι, στι 12. 5 Ιουνίου το μεσημέρι. Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Για την έκθεση Τσίκ. Τώρα, για το σημείο 7 έχει γίνει μια ανταλλαγή απόψεων τον Απρίλιο. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Σάντσε Πρεσέδο θα μας παρουσιάσει την, το σχέδιο έκθεσης. Και για αυτήν την έκθεση η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 5η Ιουνίου το μεσημέρι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Έχει ήδη γίνει ανταλλαγή απόψεων για τα βασικά σημεία του θέματος από την τελευταία μας συνεδρίαση ε, εγώ είχα την ευκαιρία να έρθω σε επαφή με την νομική υπηρεσία συζητήσαμε κάποια συγκεκριμένα θέματα, κάποιες πτυχές αυτής της έκθεσης και προσπάθησα να ε, στα έξι μία της να συμπεριλάβω τα βασικά συμπεράσματα που προέκυψαν. Δεν θα επαναλάβω τόσο είπαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση. Απλά να σας πω ότι με τη νέα συνθήκη της Λισαβόνας στο άρθρο 290 ε, και στο άρθρο 291 καθορίζονται οι κατεξιότητες πράξεις και οι εκτελεστικές πράξεις. Πρόκειται για μια καινούρια ε, δομή ε, της ιεραρχίας των νομικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παλιότερα υπήρχαν μόνο οι εφαρμοστικές πράξεις, τώρα έχουμε και τις πράξεις κατεξιοδότηση με πολύ συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και με παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η απόφαση του ε, πότε θα πρέπει να εκδίδονται οι μεν και πότε οι δε είναι πολιτικής φύσεως κυρίως, αλλά ε, θα πρέπει να ε, υφίστανται, μια νέα σειρά κριτηρίων που θα καθορίζουν το πώς θα λαμβάνεται αυτή η απόφαση. Θέλουμε να εξασφαλίσουμε και καλή ποιότητα στην νομοθεσία και επαρκή έλεγχο από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ένα άλλο θέμα είναι η, εφα, η e προσαρμογή των παλιότερων διαδικασιών που υπήρχαν στις, στα καινούργια δεδομένα της συνθήκης της Λισαβόνας. Σε ό,τι αφορά την αλληλεία, την αλληλεία είχαμε την διαδικασία με έλεγχο και δεν νομίζω ότι θα μας δημιουργηθούν ιδιαίτερα προβλήματα για την προσαρμογή της. Να σας ε, μιλήσω για τα διάφορα θέματα τα οποία προτείνω να συμπεριλάβουμε στην έκθεση. Θα ήθελα να ακούσω την τοποθέτηση των συναδέλφων προκειμένου να λάβω υπόψη τις απόψεις τους. Πρώτο θέμα, η επιλογή του κατάλληλου νομοθετικού μέσου νομικού μέσου μάλλον, δεν είναι ε, τεχνικής φύσεως αλλά πολιτικής φύσεως. Οι νομοθετικές ε, πράξεις θα πρέπει να περιλαμβάνουν τα βασικά σημεία. Βασικά σημεία τα οποία ε, δεν μπορούν να εκχωρηθούν, είναι αρμοδιότητα του νομοθέτη και δεν μπορούν να εκχωρηθούν. Πρόκειται για πολιτικές πτυχές, οικονομικούς στόχους που άπτονται των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών μας λοιπά Αυτά τα βασικά στοιχεία και ο αποτελεσματικός έλεγχος θα πρέπει να παραμείνουν προφανώς στα χέρια του νομοθέτη. Το νομικό μέσο που θα επιλεγεί είναι σημαντικό και για την ισορροπία μεταξύ των εξουσιών και για τη βελτίωση της ποιότητας του νομοθετικού έργου. Πρώτο σημείο της έκθεσης αφορά λοιπόν αυτό το θέμα. Δεύτερον, υπογραμμίζω την σημασία συνέπειας, συνέπειας στην επιλογή, στην οποιαδήποτε επιλογή γίνεται. Συμφωνούμε με τη διάσκεψη των Πρόεδρων ε, που επιθυμεί ε, να λαμβάνει τις αποφάσεις αυτές με βάση κοινά κριτήρια ε, έτσι ώστε να εξασφαλίσουμε αυτή την συνέπεια στην επιλογή του κατάλληλου νομικού μέσου οχήματος. Το Κοινοβούλιο αποκτά εμπειρία σιγά σιγά σε όλα αυτά τα θέματα και με βάση αυτή την εμπειρία μπορούμε να καταρτήσουμε, να ε, υιοθετήσουμε ένα σύστημα το οποίο θα διευκολύνει το συντονισμό και την παρακολούθηση με τρόπο πιο διαρθρωμένο. Τρίτο σημείο ε, αναφέρεται στο εξής. Όπως υπάρχει ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων των διαφόρων επιτροπών στο Κοινοβούλιο, θα ήταν ενδιαφέρον να υφίσταται και ένα πολιτικό δίκτυο ο πρόεδρος για παράδειγμα της κάθε επιτροπής, ένας αντιπρόεδρος ή έστω και ένα μέλος να ε, έχει την αρμοδιότητα να συνεργάζεται με τον ομόλογο τους άλλες επιτροπές για τέτοιου είδους ζητήματα. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα αναλαμβάνει αυτό το συγκεκριμένο μέλος όλη την ευθύνη. Η δική μου ιδέα είναι ο εισηγητής κάθε έκθεσης να ενημερώνει και για την παρακολούθηση και για τη συνέχεια που δίδεται στο, στο, στο συγκεκριμένο ζήτημα. Νομίζω ότι με αυτόν τον ε, τρόπο θα ε, βελτιώνεται η εμπειρία του Κοινοβουλίου και η μελλοντική του δράση. Επόμενο σημείο της έκθεσής μου έχει σχέση με τα προβλήματα τα οποία παρουσιάστηκαν σε ό,τι αφορά την προσαρμογή της παλιότερης νομοθεσίας στα δεδομένα της Λισαβόνας. Μερικές φορές το Κοινοβούλιο, Κομισιόν και το Συμβούλιο ε, δεν επιλέγουν το κατάλληλο νομικό μέσο με τον ίδιο τρόπο με τα διακριτήρια. Πολλές φορές το Συμβούλιο ε, τίνει ε, να δίνει περισσότερο βάρος στις εφαρμοστικές πράξεις από ό,τι στις ε, κατεξιοδότηση πράξης. Γιατί με αυτόν τον τρόπο θεωρεί ότι ελέγχει καλύτερα τη διαδικασία. Τέτοιου είδου θέματα θα πρέπει να τα εξετάζει και το Κοινοβούλιο. Το Κοινοβούλιο δεν θα πρέπει να χάσει τη δυνατότητα ελέγχου, την εξουσία ελέγχου που του δίδεται. Δεδομένου το άρθρο 290 καθορίζει τους όρους για την εκχώρηση αρμοδιοτήτων, θα μπορούσαμε ε, να επιλέξουμε κάποια κριτήρια πιο ουδέτερα έτσι ώστε το Συμβούλιο να μην επιλέγει ε, ε, τόσο συχνά τις εφαρμοστικές πράξεις που αποδίδουν στο Κοινοβούλιο μικρότερο, λιγότερο σημαντικό ρόλο ελέγχου. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε μια κατάλληλη μέθοδο για την χρήση αυτών των διαδικασιών. Επόμενο σημείο αναφέρεται στην ε, λισβονοποίηση, λισαβονοποίηση, ε, στην προσαρμογή δηλαδή στα δομένα της Λισαβόνας. Αυτή η διαδικασία θα πρέπει να ε, ολοκληρωθεί με το τέλος της ε, θητείας μας. Δηλαδή θα πρέπει να έχουμε, την έχουμε ολοκληρώσει του χρόνου πριν γίνουν οι επόμενες ε, Νομίζω ότι μία θητεία μας είναι επαρκής για την προσαρμογή στα δεδομένα της συνθήκης Λισαβόνας. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο θα έπρεπε να στείλουμε. Ενώ στο σημείο 6 προτείνουμε να καταλήξουμε σε μια κοινή συμφωνία με το Συμβούλιο και την Κομισιόν για την ερμηνεία αυτών των άρθρων της Συνθήκης Λισαβόνας ε, και την παρακολούθηση της εφαρμογής τους. Αυτές είναι οι θέσεις μου και θα ήθελα να ακούσω την άποψή σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Σάντσες Πρεσέδο. Δεν έχει ζητήσει κάποιος το λόγο. Η κυρία Τομάς. Ναι, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Συμφωνώ απολύτως με την άποψη και τα επιχειρήματα του κυρίου Σάντσες Πρεσέδο. Θα ήθελα απλώς να προσθέσω μία ανησυχία για την πτυχή της ευθύνης του Κοινοβουλίου. Και εδώ συμφωνώ με τον κύριο Σάντσες ε, Πρεσέδο. Ο νομοθέτης δεν θα πρέπει να αποποιείται των ευθυνών του ε, όταν πρόκειται ιδέως για νομοθετικές πράξεις. Προσωπικός, ε, στη συγκεκριμένη περίπτωση και μάλιστα ασχολήθηκα και με το θέμα αυτό για την εφαρμογή των όρων της Λισαβόνας στον ε, κανονισμό ε, πώς θα μπορέσει στην πραγματικότητα να ελέγξει το Κοινοβούλιο της πράξης κατά εξονσιοδότηση. Αυτή τη στιγμή είναι λίγες οι κατεξουσιοδότηση ε, πράξεις, διότι δεν έχουμε φτάσει στο απόγειο της εφαρμογής. Υπάρχουν ακόμα κάποιοι κατάλογοι που έρχονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ε, οι οποίοι είναι αρκετά ουσιαστικοί. δεν μπορούμε ακόμα να ξεκινήσουμε μια διαδικασία ελέγχου, αλλά θα υπάρξει ένας κοινοβουλευτικός έλεγχος με την ευθύνη του Κοινοβουλίου, η οποία ε, θα περιλαμβάνεται μεν ε, θα υπάρχει και εγγράφος, αλλά στις πράξεις κατεξουσιοδότηση στη συνέχεια δεν θα υπάρχει κανένας έλεγχος δεν ξέρω αν βρεθούμε ενώπιον μιας κατάστασης ε, ώστε να χρειαστεί στη συνέχεια να λάβουμε μέτρα. Ε, είμαστε υπεύθυνοι και αναλαμβάνουμε μια ευθύνη χωρίς να έχουμε μια πραγματική στην πραγματικότητα δυνατότητα να ελέγξουμε την κατάσταση εάν αρχίσουμε αυτή τη διαδικασία. Ευχαριστώ. Ναι, κάποιος άλλος θέλει το λόγο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. κανείς. Κύριε Σάντσες Πρεσέδο, ναι, θα ήθελα να ευχαριστήσω την συνάδελφο, την κυρία Τομάς, για την παρέμβασή της. Είναι προφανές, είναι δύο πτυχές τις οποίες συζητάμε. Καταρχάς ε, η δημοκρατική αρχή αφενός, δηλαδή η νομιμότητα των αποφάσεων που εγκρίνονται και από εκεί και πέρα η αποτελεσματικότητα της δημοκρατίας. Αυτές είναι δύο ε, ουσιαστικές πτυχές ε, της ζωής των θεσμικών οργάνων. Ο νομοθέτης προφανώς και θα πρέπει να διατηρήσει τα ουσιαστικά στοιχεία και για τον ίδιο. Αυτά ε, δεν μπορεί να τα, τα βάσει σε κανέναν. Υπάρχει και μία απόφαση του δικαστηρίου που εμένα μου φαίνεται πολύ ενδιαφέρουσα, 5 Σεπτεμβρίου του 2012 και λέει ότι οι πολιτικές αποφάσεις προποθέτουν ότι ε, συγκλίνουν διστάμενες απόψεις επί τη βάση συγκεκριμένη νομοθεσία. Εδώ υπάρχει συγκεκριμένη πολιτική εκτίμηση που λέει ότι ο νομοθέτης είναι αυτός ο οποίος πρέπει να υλοποιήσει και υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία χαρακτηρίζουν τις πολιτικές αποφάσεις που είναι αποφάσεις που αφορούν κυρίως θεμελιώδη δικαιώματα ή ε, με σκοπό συγκεκριμένα αποτελέσματα τα οποία αναμένουμε ή την προσφυγή σε συγκεκριμένους πόρους. Αυτά είναι τα βασικά στοιχεία. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι ο νομοθέτης ε, δεν μπορεί να διατηρήσει κάποια στοιχεία και για τον εαυτό του, όλα τα στοιχεία τα οποία θεωρεί σημαντικά προκειμένου να καταλήξει σε κάποιο πολιτικό αποτέλεσμα, θα μπορούσε και αυτά να τα διατηρήσει για τον ίδιο. Ε, ακόμα και αν δεν είναι τόσο ουσιαστικά. Και επίση ο νομοθέτη θα πρέπει να διασφαλίσει ότι είναι αποτελεσματική η νομοθεσία του. Επομένω, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ε, προποθέτει και μηχανισμού ελέγχου και παρακολούθηση, ώστε οι εντολέ του να τηρούνται και να είναι αποτελεσματικέ. Αυτό είναι θέμα ποιότητα τη δημοκρατία και επομένως θα πρέπει ε, αυτά τα οποία έχουν κατά νου να μεταφράζονται σε πραγματικότητα στην καθημερινή μας ζωή. Δεν είναι απλώς ε, λοιπόν για η δημοκρατία, θα πρέπει να έχει και αποτελέσματα για τους πολίτες μας. Και ευχαριστώ πολύ λοιπόν την κυρία Τομάς για την παρέμβασή της και ε, κάποια νοήματα που μου έκανε η κυρία Φράγα. Είμαι εν αναμονή των τροπολογιών σας και ελπίζω να μπορέσω να τις συμπεριλάβω ε, στην έκθεση και αν χρειαστεί να διορθώσω και την έκθεση για να λάβουμε υπόψη και τις θέσεις σας. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Αν δεν υπάρχει κάποια άλλη παρέμβαση, να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ενημέρωση για την αντιπροσωπεία στις Κανάριες νήσιους. Ε, έξι συνάδελφοι είχαμε πάει στις Κανάριες νήσους και θα υπάρξει και μία συνολική έκθεση για την επίσκεψη, αλλά εγώ θα σας κάνω μία περίληψη. Τα έχετε όλα στην έκθεση. Η, έκθεση, η επίσκεψη συγγνώμη, έγινε καταρχάς ε, προκειμένου να επισκεφθούμε το κέντρο ελέγχου. Ακούστηκαν όχι μόνο πολλές φήμες, αλλά και πολλές και διαφορετικές ερμηνείες και ανακοινώσεις για τη δυνατότητα που είχε το λιμάνι στη Λασπάσμας να ελέγξει τις εκφορτώσεις και αν υπήρχε ένα κατάλληλο κέντρο ελέγχου. Υπήρχε και ένα άλλο ε, σημείο το οποίο ήταν σημαντικό για τις Καναρίες νήσους αλλά και για την Ισπανία. Ε, η παρούσα κατάσταση των αλευτικών συμφωνιών με το Μαρόκο και τη Μαυρτανία. Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν πολύ στα θέματα αυτά την διάρκεια της πρώτης ημέρας ήταν ε, ε, συνεχής η επίσκεψη. Όλη μέρα ήμασταν στο λιμάνι του Λασπάλμας από το πρωί μέχρι το βράδυ και ε, συναντηθήκαμε στην πραγματικότητα με όλους τους ενδιαφερομένους. Ήταν και ο επικεφαλής της λιμενικής αρχής εκεί, αλλά φυσικά και με αλληλείς και με συνδικάτα, με κυβερνητικές οργανώσεις, το σύνολο του ελευτικού κλάδου και με πολιτικές αρχές παρουσιάστηκε μια γενική εικόνα του λιμένα. Δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στο θέμα του ελέγχου της αλληλείας και νομίζω ότι από αυτά μείναμε πάρα πολύ καλοί ικανοποιημένοι και διαπιστώσαμε ότι ο λιμένας αυτός αποτελεί πλέον πρότυπο το οποίο θα πρέπει να ακολουθούν και άλλοι λιμένες τους οποίους ε, δεν ακολουθούνται οι ίδιες διαδικασίες ελέγχων ε, για τα ε, αλληλεία. Ε, την πρώτη μέρα επικεντρωθήκαμε επίσης ε, στις ε, αγροοικονομικές συνέπειες των συμφωνιών ελευθέρου εγκουμπορίου και των συμφωνιών πιο συγκεκριμένα της Μαυριτανίας και του Μαρόκου. Ε, κατέστη σαφές ότι υπάρχει ανησυχία για την συμφωνία και το μήνυμα είναι ότι για τη συμφωνία για τη Μαυριτανία ειδικά θεωρείται ότι δεν είναι βιώσιμη. Τα σκάφη είναι δεμένα στα λιμάνια χωρίς δυνατότητα αλληλείας και οι άδειε αλήψεις δεν χρησιμοποιούνται. Την επόμενη μέρα επισκεφτήκαμε το Λανθαρότε. Είδαμε κάποιες ε, ηχθειοκαλλιέργειες, ε, τις ε, σημαντικότερες εκμεταλλεύσεις ηχθειοκαλλιέργειας των Καναρίων νήσων και της Ισπανίας. Και στη συνέχεια επισκεφθήκαμε ένα εργοστάσιο μεταποίησης. Το ταξίδι λοιπόν ήταν πλήρες μάθαμε τα πάντα, από το τι κάνουν τα ψάρια στη θάλασσα μέχρι το πώς ε, φτάνουν σε κονσέρβες και κουτιά για την ε, εμπορία τους. Και μιλήσαμε φυσικά και με κάποιους αλληλείς, εκπροσώπους ερασιτεχνικής αλληλείας, οι οποίοι ε, μας ανέφεραν την ανησυχία τους για τον ορισμό της ερασιτεχνικής αλληλείας, αλλά και το τι θα γίνει με τη μεταρρύθμιση και τι θα γίνει με αυτούς στη διάρκεια της μεταρρύθμισης. Και τέλος, συνεδριάσαμε με τον τομέα των κεφαλόποδων που ε, ενδιαφέρονται ιδιαίτερα για τη συμφωνία με τη Μαυρτανία. Ήταν τρει πλήρε μέρες, ε, ο ήλιος δεν μας είδε καθόλου, όχι μόνο γιατί δεν βγήκαμε καθόλου στην Ήπεθρο, στα Γανάρια νησιά, αλλά γιατί είχε και κακοκαιρία. Ε, ίσως αν υπήρχε ο ήλιος ε, θα νιώθαμε καλύτερα να είμαστε εκεί, να απολαύσουμε τον καλό καιρό και τελικώς απλώς χρειάστηκε να δουλεύουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτοί οι οποίοι ίσον βίωσαν την εμπειρία. Η κυρία Ρόντουστη ήταν εκεί, δεν βλέπω κάποιον άλλον εδώ στην αίθουσα, αλλά έχετε και την έκθεση. Αν θέλετε οποιαδήποτε διευκρίνηση, είμαι στη διάθεσή σας και θα ήθελα να ευχαριστήσω και όλους όσους ήταν εκεί για το καλό πνεύμα συνεργασίας, ε, κάτι το οποίο φυσικά ε, ισχύει εδώ και ε, μας ενδιαφέρει ιδιαίτερα για όλους όσους ε, συναντήσαμε εκεί και κυρίως ε, τη Λιμενική Αρχή. Κυρία Ρόντουστη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω θερμά. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον ταξίδι, ιδιαίτερα όσον αφορά τη Μαυριτανία. Σήμερα θα ψηφίσουμε σχετικά με το θέμα αυτό. Λάβαμε πάρα πολλές πληροφορίες και θα ήθελα προσωπικά να σας ευχαριστήσω για το εξαιρετικό πρόγραμμα. Να συστήσω σε όλους ε, να επισκεφτούν τα Καράρια. Έχουμε να μάθουμε πολλά εκεί και είναι και υπέροχα νησιά. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ κύριε για την σύστασή σας. Άλλα θέματα σταματάμε και ξαναρχίζουμε στις 3 με τις κάρτες σας για τις πιοφορίες.